Ladies and gentlemen, a warm welcome. Και κύριοι, σας καλωσορίζω θερμά στη διάσκεψή μας για το μέλλον των ε, αποστολών παρατήρηση εκλογών. Είναι καταπληκτικό που η αίθουσα είναι γεμάτη με τόσους πολλούς συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Πριν ξεκινήσουμε σας παρακαλώ να δούμε ένα σύντομο βίντεο για τις αποστολές παρατήρησης ε, της Ένωσης ως εισαγωγή. Παρακαλώ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 Σας ευχαριστώ για αυτό το θαυμάσιο βίντεο, κύριε και κύριοι. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε διερμηνία από και προς αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και ελληνικά. Παρακαλώ, ε, κοιτάξτε τις ε, καμπίνες για να δείτε τον αριθμό της γλώσσας, αν θέλετε. Ε, πρόκειται να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη. Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμη. Ε, έχει άλλες σημαντικές δεσμεύσεις, υποσχέθηκε ότι θα έρθει αργότερα. Να ξεκινήσω λοιπόν ε, καλωσορίζοντάς σας τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλους τους άλλους μας προσκεκλημένους. Είναι μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω σε αυτήν την διάσκεψη υψηλού επίπεδου που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση με τη στήριξη τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό που είστε τόσο πολύ εδώ παρόντες, ότι δηλαδή υπάρχει τόσο ευρύ ενδιαφέρον από τόσο πολλές χώρες για αυτήν την συνδιάσκεψη. Δίπλα μου είναι ο συνάδελφός μου κύριος Αντώνιο Παντσέρη, που είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπινών Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ λέγομαι David McAllister. είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και μαζί θα προεδρεύσουμε σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση. Τώρα, μερικά λόγια για μένα. Από μένα μάλλον, για το τι κάνουμε εμείς ε, σε αυτό το τομέα. Από ό,τι θα ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το άμεσα εκλεγμένο κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη 751 ως μέλη. Είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο στον κόσμο μετά το Κοινοβούλιο της Ινδίας και το μεγαλύτερο διεθνικό δημοκρατικό κοινοβούλιο στον κόσμο. Γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά όλοι τις εκλογές, τις εκλογικές διαδικασίες. Έχουμε ποικίλε εμπειρίες με εκλογικά συστήματα, με ενδεχόμενα νοθείας και άλλες ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει κανείς εκλογές. Και έχουμε ξεκινήσει την προπαρασκευή για το μεγαλύτερο εκλογικό γεγονός στην Ευρώπη που λαμβάνει η χώρα κάθε πέντε χρόνια, τις δικές μας εκλογές. Τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα γίνουν τέλη Μαΐου του 19. Είμαστε λοιπόν σε προεκλογικό κλίμα και γι' αυτό ε, είναι μεγάλη τιμή που έχουμε αυτήν τη τόσο σημαντική και επίκαιρη εκδήλωση για την παρατήρηση των εκλογών παντού στον κόσμο. Θέλω να τονίσω ότι η πρόθεση τη δημοκρατία, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη καλή διακυβέρνηση είναι η ουσία τη ταυτότητα τη Ένωση και αναφέρονται σε όλα τα ιδρυτικά κείμενα και του βασικού στόχου τη πολιτική μα εξωτερικών και ασφάλεια. Οι εκλογέ είναι ουσιώδε βήμα στην οδό προ τη δημοκρατία. Είναι το μέσο για να υπάρξει πολιτική συμμετοχή των πολιτών και αναγκαίο στοιχείο για την πλήρη άσκηση μια σειρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη στην υποστήριξη εκλογικών διαδικασιών ε, παντού στον κόσμο, όπω έδειξε και το βίντεο, μέσω τη ανάπτυξη ε, τη λειτουργία διαφόρων φορέων διαχείριση των εκλογών, μέσω προγραμμάτων ε, αγωγή των πολιτών και εκλογέων και μέσω των αποστολών παρατήρηση. Δυστυχώ, η στόχη, η μεθοδολογία και οι βασικέ αρχέ των παρατηρήσεων εκλογών μπορεί να παρανοηθούν από ορισμένου, από ορισμένα μέσα και από ορισμένε αρχέ και μπορεί να οδηγήσουν σε επικρίσει και η πίεση επί των παρατηρητών αυξάνει και μάλιστα ταχαίω. Οι παρατηρητέ εκλογέ πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτέ τι ε, προκλήσει για τι σύγχρονε εκλογέ, ιδιαίτερα λόγω της χρήσης της ε, τεχνολογίας, της πληροφορίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και επιπλέον υπάρχει δυνατότητα εξωτερικού επηρεασμού που μπορεί να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η διάσκεψη σήμερα και αύριο ελπίζουμε ότι θα μας δώσει σε όλους ε, μέλη του Κοινοβουλίου, επικεφαλής ε, εκλογικών φορέων, εκλογικών επιτροπών, καθώς και άλλων εμπειρογνωμόνων και εκπροσωπών των ε, οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών να αντιμετωπίσουμε όλε τι προκλήσει και να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε καλύτερα τι ε, παρατηρήσει εκλογών στι συνθήκε του 21ου αιώνα. Και δεν μιλάω μόνο θεωρητικά. Ο κ. Παντζέρη, αλλά και εγώ, όπω και πολλοί άλλοι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι εδώ παρούσε και παρόντε, στα πρώτα έδρανα, έχουμε όλοι διαπιστώσει τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι παρατηρητέ εκλογών. Εγώ ήμουν ε, επικεφαλή τη Αποστολή παρατήρησης του 2017 στην Κένια. Και θυμάστε πόσο μεγάλα ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Και η περίπτωση του Γκαμπών επίση ήταν πολύ δύσκολη αποστολή και είμαι σίγουρο ότι η Επίτροπο Γκάμπριελ που είναι εδώ δίπλα θα σα εξηγήσει περαιτέρω. Και καλωσορίζω και την ε, Επίτροπο. Είναι τιμή που σας έχουμε μαζί μας. Και ε, όπως ε, ήδη είπα, οι περισσότεροι συνάδελφοι σε αυτή την αίθουσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε έχουν προεδρεύσει είτε έχουν συμμετάσχει σε αποστολέ παρατήρηση ή έχουν συμμετάσχει σε αποστολέ ε, παρατήρηση που έχει οργανώσει η Ένωση ή οι οργανισμοί των Ηνωμένων και του ε, ΟΑΣΕ. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει εδώ και πάνω από 30 χρόνια σε αποστολέ παρατήρηση εκλογών. Έχουμε ένα ειδικό σώμα για αυτές τις παρατηρήσεις. Είναι η λεγόμενη ομάδα συντονισμού για τις εκλογές. Είναι γνωστή ως DEG που και συμπροεδρεύεται από την Λίντα Μακάβαν που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και από εμένα. Συντονίζουμε έτσι όλες τις δραστηριότητες παρατήρησης των εκλογών τους ώστε να υπάρχει μια συνέπεια και δίνει συμβουλές στην κυρία Μογκερίνη για τις προτεραιότητές μας όταν παρατηρούμε εκλογές. Και η πείρα μας δείχνει ότι έχει αποδείξει ότι έχει σημασία για την ε, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ε, προσπάθεια εντοπισμού και ε, διεξαγωγής τέτοιων αποστολών. Πιστεύω και ελπίζω ότι όλοι, όλα τα κοινοβούλια που συμμετέχουν στην σε αποστολές παρατήρησης αναγνωρίζουν την σημασία Δημιουργία στη χώρα του ενό παρόμοιου σώματος. Να δώσω το λόγο στην ε, Μαρία Γκάμπλ που είναι επίτροπο για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία. Έχει μεγάλη πείρα, έχει συμμετάσχει σε εκλογέ και στην ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στο Γκαμπόν. Έχετε πάει σε πολλά μέρη Μαρία κατά την ε, θητεία σα. Έχετε πάει στο Τόκο, το Γυργιστάν, την Τανζανία, το Σουδάν, το Τσάτ, την Αιγυρία, τη Σιέρα Λεόν, την Μπουρκίνα Φάσο, την Ουγγάντα και την Ιορδανία. Και ορισμένε φορές προλάβατε να είστε και εδώ στι Βρυξέλλε. Εντυπωσιακός κατάλληλο χωρών, πολύ έντονη πείρα παρατήρηση εκλογών. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς που εργαζόμαστε στις ε, εξωτερικές σχέσεις ε, ε, μας λείπετε. Μαρία, να σου δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Ντέιβιτ, κύριε Παντζέρη, αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συμμετέχοντες στη διάσκεψη, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την χαρά μου και την ικανοποίησή μου που βρίσκομαι ενώπιόν σας και βλέπω και όλα αυτά τα πρόσωπα που δεν είναι απλώς γνωστά επειδή ήμασταν συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και επειδή ε, ζήσαμε πολλά ε, μαζί επί τόπου. Και ναι, Ντέιβιτ, εάν ε, όλη αυτή η εμπειρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και την παρατήρηση εκλογών και όλοι αυτοί οι αγώνες σε φέρουν στα ψηλά αξιώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας εύχομαι και εσείς να περνάτε λίγο χρόνο στις Βρυξέλλες. Το θέμα μας είναι οι αποστολές παρατήρησης εκλογών. Είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο ε, πολύτιμο και απαράμιλο για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την υποστήριξη της δημοκρατίας και ε, της αξίας μας, που είναι προσφυλής σε όλους. Και πέρα από κάθε ρομαντική διάθεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποστολή να φροντίζει εκλογές να είναι χωρίς αποκλεισμούς δίκαιες, διαφανείς και δημοκρατικές παντού, σε όλο τον κόσμο. Παρ' αυτά γνωρίζουμε ότι για να υπάρξει μια διεθνής ακτινοβολία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή θα πρέπει να εγγράφεται στην προάσπιση των δημοκρατικών αρχών και αξιών μας, τη διαρκή και μόνιμη. Δεν είναι καθόλου και εκτιμένο αυτό. Για μας, η δύναμη μας είναι να τα διατρανώνουμε όλα αυτά. Η ελευθερία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία είναι αδιαπραγμάτευτα. Ε, είναι γενή δικαιώματα για κάθε άνθρωπο και εμεί οι Ευρωπαίοι συνεργαζόμαστε με την Αφρικανική Ένωση, με τα Ηνωμένα Έθνη και είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες και έξω από τα σύνορά μας καμιά φορά. Πιο συγκεκριμένα οι αποστολέ παρατήρησης εκλογών είναι ένα πολύ προβεβλημένο μέσο, πολύ αποτελεσματικό και ε, γνωστό. Γιατί Α μην είμαστε αφελεί. Υπάρχουν κάποιε άλλε δυνάμει που δεν έχουν την ίδια θεώρηση για τα πράγματα στον κόσμο με εμά και προσπαθούν να αυξήσουν την επιρροή του. Και ένα από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν είναι η χειραγώγηση των εκλογών για να φτάσουν στου στόχου του. Παρ' όλα αυτά, πριν περάσω στις προκλήσεις για τις εκλογές και τις αποστολές παρατήρησης εκλογών που απορρέουν από την ψηφιακή εποχή, θα ήθελα λίγο να επιμείνω στα δυνατά μας σημεία. Οι αποστολέ παρατήρηση εκλογών σημαίνουν ε, περάσπιση των δημοκρατικών αρχών και αξιών μα και ε, διαφύλαξη τη ακαιρεότητα εκλογική αναμέτρηση. Και αυτή είναι η ισχύ και η δύναμή μα. Βασιζόμαστε στην ανεξαρτησία. Δεν είναι τυχαίο που ηγείται πάντα κάποιο πολιτικό, ένα ευρωβουλευτή σε αυτέ τι αποστολέ παρατήρηση εκλογών, που είναι επικεφαλή, ακριβώ για να μπορέσει να υπερασπιστεί αυτή την πολιτική του ανεξαρτησία. Η άλλη δύναμή μας είναι η μεθοδολογία μας που είναι πάρα πολύ αυστηρή. Το είδαμε και κατά ε, τη διάρκεια του βίντεο. Πάντα έχουμε αξίες και ε, κώδικες που θέλουμε να μοιραζόμαστε με όσο γίνεται περισσότερος ακριβώς ε, όταν έρχεται η ώρα της αξιολόγησης θα πρέπει να έχουμε κοινού κανόνες και πρότυπα. Και η τρίτη μας δύναμη και είναι η συνεργασία με άλλες αποστολές παρατήρησης εκλογών. Πόσες φορές δεν είδαμε επί τόπου πόσο σημαντικό είναι να ε, μπορείς να συντονίζεσαι με κάποιο άλλο. Έτσι και από πλευράς επιμελητίας για να καλύπτουμε όσο γίνεται περισσότερες περιφέρειες. Ξέρουμε ότι όλοι έχουμε περιορισμένους πόρους και ανθρώπινους και οικονομικούς. Και είναι πολύτιμο να μπορείς να ανταλλάσσεις πληροφορίες στη συνέχεια και όταν κάνουμε την προκαταρκτική δήλωση να μπορούμε όλοι να μιλούμε με μία φωνή, γιατί στο κάτω-κάτω αυτή είναι η φωνή της δημοκρατίας, του κατευνασμού, της προστασίας ε, των δικαιωμάτων των πολιτών που εκφράζεται. Και περνώ αμέσω στις νέες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώνετε τόσο μεγάλο χρόνο φέτος στο θέμα αυτό. Μάλιστα, σήμερα η παρατήρηση εκλογών αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις και νομίζω ότι θα ήταν σωστό να πούμε ότι αντανακλούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες μας και η κυριότητά τους. Παραπληροφόρηση, στοχευμένες εκστρατείες ε, στα ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι νέες τεχνολογίες είναι εκείνες που μπορούν να έχουν και πάρα πολύ θετικές επιπτώσεις, αλλά έχουν και κινδύνους και μπορούν να έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες κατά τον τρόπο αυτό. Ως καλή λοιπόν επικεφαλής παρατήρησης εκλογών, όταν εκλήθη να εξετάσω αυτά τα θέματα, ε, σκέφτηκα τις τρεις φάσεις. Τι γίνεται πριν την εγγραφή των ε, ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους, τι γίνεται τη μέρα των εκλογών και τι γίνεται μετά τις εκλογές, όταν ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα. Προφανώς αυτά τα τρία στάδια μπορούν να έχουν περισσότερη διαφάνεια με τις νέες τεχνολογίες, μεγαλύτερη κινητοποίηση των ψηφοφόρων ή ακόμα και πρόσβαση σε ένα γενές δικαίωμα κάθε πολίτη το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα στη συμμετοχή στα κοινά. Για τον λόγο αυτό λοιπόν προβληματίστηκα πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και τις νέες πλατφόρμες για τη διοργάνωση εξτρατιών ενημέρωσης που θα φτάνουν σε πολίτες όσο γίνεται περισσότερος, τις γυναίκες, στην Ήπεθρο, στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, Σκέφτομαι εδώ την ανάγκη να ενταχθούν νέες τεχνολογίες ε, όταν εκπαιδεύουμε ε, παρατηρητές εκλογών επί τόπου. Ξέρουμε όλοι μακροπρόθεσμα ότι οργανώνεται και μια αποστολή ε, τοπική παρατήρηση εκλογών που μπορεί να διαδεχθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους οργανισμούς που κάνουν παρατήρηση εκλογών. Εδώ είναι πολλές οι προκλήσεις. Το βασικότερο είναι η κυβερνοασφάλεια. Και τώρα ακόμα. Έχουμε προγράμματα που τρέχουν. Επιτρέψτε μου να σα αναφέρω μερικά. Έχουμε στη Σενεγάλη για την καταγραφή των εκλογέων για ένα ε, εθνικό σύστημα ταυτότητας. Επίσης, ένα σύστημα καταγραφής στο Μαλί, στο Καμερούν, στο Νίγηρα, στη Σιέρα Λεόνε. Όλα αυτά τα προγράμματα τρέχουν και θα πρέπει να φροντίσουμε η κυβερνοασφάλεια να είναι αναπόσπαστο τμήμα όλης της διαδικασίας από την αρχή μέχρι το τέλος, διότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι μόνο οι ε, επιθέσεις σε σχέση με τα προσωπικά μας δεδομένα. Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν γνωρίζουν σύνορα. Αυτό μπορεί να αφορά και κρίσιμες υποδομές και κρίσιμες υποδομές είναι και οι εφορευτικές επιτροπές. Παραμένει λοιπόν μεγάλη αυτή η πρόκληση. Η εκλογική κατάλογη, οι εκλογές, τα εκλογικά τμήματα και η ε, φύλαξη των δεδομένων και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για μένα, προστασία των προσωπικών δεδομένων, για να μπορούν να προχωρήσουν οι προτάσεις. Πρέπει να βλέπουμε πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα στα δίκτυα κοινωνικής ε, μάλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς έχουμε το περίφημο GDPR, τον κανονισμό για την προστασία ε, των προσωπικών δεδομένων, το σημαντικότερο στον κόσμο. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και 53 χώρες αναπτυσσόμενες που στερούνται ε, εθνικής νομοθεσίας ή έχουν μια πλημελή ε, νομοθετική ρύθμιση για το μέλλον, για τις ε, επόμενες ευρωεκλογέ θα κάνω κάποιες προτάσεις, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα θέματα και για άλλες εκλογές. Παραμένει κομβικό όμως αυτό. Και φυσικά δεν μπορώ να παραλείψω το θέμα των ψευδών ειδήσεων, των fake news και της παραπληροφόρησης. Προσωπικά έχω αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Όταν ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, παρατήρησης εκλογών στην Καμπών. Πραγματικά ήρθαμε αντιμέτωποι με μια σημαντική εκστρατεία παραπληροφόρησης, ενορχιστρωμένη, που στρεφόταν άμεσα κατά ε, της ομάδας μου και μου προσωπικά. Σήμερα θα πρέπει περισσότερο να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Η παραπληροφόρηση βλάπτει την εμπιστοσύνη και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στα θεσμικά όργανα και ο ένας τον άλλον. Και μετά το σκάνδαλο της Cambridge Analytica γνωρίζουμε πολύ πόσο οι καμπάνιες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα εκείνους οι οποίοι αποτελούν το κεντρικό και το σημαντικότερο στοιχείο κάθε εκλογής, δηλαδή με τα λόγου γνώσεως να επιλέγει ο πολίτης τι θα ψηφίσει για να το κάνει αυτό, θα πρέπει η πληροφόρηση να μπορεί να διασταυρώνεται και να ενημερώνεται σωστά και δημόσια ο πολίτης. Εργαζόμαστε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Δεν υπάρχουν πανάκες και θαυματουργές λύσεις, αλλά χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση, στην πολιτική προβολή. Για τη διαφάνεια των αλγορίθμων γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα μπορούν να επηρεάσουν την αίσθηση που έχουμε για την πραγματικότητα. Και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο μπορούμε να μεταφέρουμε αυτές τις εμπειρίες. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στη ρητορική μίσους, hate speech. Αυτό συνδέεται με τις βίες εκφράσεις στις εκλογές. Η βία δεν είναι μόνο σωματική βία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα εθελοντικό κώδικα διοντολογίας. Θα μπορούσαμε όμως να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το θέμα για να το μεταφέρουμε και σε άλλα πλαίσια, στην προεκλογική εκστρατεία. Να δεσμεύονται οι βασικότεροι υποψήφοι για να κατευνάσουν τα, τα πνεύματα. Γνωρίζουμε πόσο αυτό μπορεί να έχει ανετικές επιπτώσεις και πραγματικά ε, με ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό. Θα ήθελα επίσης να επιμείνω στο θέμα των νέων τεχνολογιών και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια. Όλο και περισσότερο ε, σκέφτομαι και τη τεχνολογία blockchain ε, που έχει μεγαλύτερη ιχνηλασιμότητα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια κρίσιμη φάση. Όταν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στο εκλογικό τμήμα, θα πρέπει οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη ότι αυτά τα αποτελέσματα θα φτάσουν ε, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, τα συγκεντρωτικά και θα είναι τα σωστά. Χάρη στις νέες τεχνολογίες μπορούμε να ενισχύσουμε και την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια και να διαφυλάξουμε την ακαιρεότητα της εκλογικής αναμέτρησης. Έτσι ε, θα προάγονται οι δημοκρατικές αξίες. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε προτείνει κάποια συγκεκριμένα μέτρα για τις επόμενες ευρωεκλογέ. Εδώ και τρεις εβδομάδες έχουμε απευθύνει συστάσεις για τις επόμενες ευρωεκλογέ. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και να εστιάσουμε στη συνεργασία των ε, Εθνικών Εφορευτικών Επιτροπών με τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σήμερα επιμένουμε στη διαφάνεια. Οι πολίτες και οι ψηφοφόροι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιος χρησιμοποιεί τα δεδομένα τους, πώς τα χρησιμοποιεί και για ποιο σκοπό. Πολλό δε μάλλον που κατά τη διάρκεια μιας εκλογικής αναμέτρησης μπορεί να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Και πάλι θέλουμε να είναι διαφανής η πολιτική διαφήμιση, να γνωρίζουμε δηλαδή ποιος χρηματοδοτεί ένα περιεχόμενο ε, διαφήμισης, για ποιο λόγο, για να μπορούμε να επιλέγουμε και να αποφασίσουμε ως πολίτες με τα λόγου γνώσεως. για τα θέματα που κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι οι νέες τεχνολογίες είναι ευκαιρία πραγματική. Έτσι ώστε να επικρατήσει αυτή η διαφάνεια που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και στην εκλογική διαδικασία και στη δημοκρατία. Βέβαια συνοδεύονται και από κινδύνους οι ευκαιρίες αυτές. Αλλά αυτό λύνεται μόνο με συνεργασία, μόνο αν απευθυνόμαστε άμεσα στους πολίτες, με συγκεκριμένα μέτρα, χωρίς να θέλουμε να βρούμε λύση για όλα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις νέες αυτές προκλήσεις. Και αυτές οι προκλήσεις δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε για το μέλλον. Είναι εδώ, είναι παρούσες και χρειάζονται σήμερα απαντήσεις. Και για το λόγο αυτό σας συγχαίρω για άλλη μια φορά ε, που επιλέξατε τα θέματα για το συγκεκριμένο πάνελ ε, φέτος. Δεν θέλετε να κάνετε διαπιστώσεις, απαντήσεις θέλετε να βρείτε. Για όλα αυτά που σας παρουσίασα δεν είναι κάτι το μοιραίο. Είναι μια ευκαιρία και από κοινού θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με συνέργειες, με συνεργασίες και έτσι θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών με σθένος και στα λόγια και στις πράξεις μας για να ενισχύσουμε τις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Αυτός είναι ο δρόμος και δεν θα αλλάξει τίποτα η ψηφιακή εποχή. Και αυτό θα το αποδείξουμε με τη δύναμη του ανθρώπου. Ποτέ δεν πρόκειται οι μηχανές και τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τη δημιουργικότητά μας, ε, τις ε, κοινωνικές σχέσεις, ε, τα συναισθήματα και τις αξίες και τις αρχές. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε τόσο πολύ και με τέτοια θέληση να προωθήσουμε αυτό το κοινό μας μέλημα. Maria Gabriel, Commissioner. Αγαπητή Μαρία, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Είναι πραγματικά πολύ ε, ευχάριστο να σας ακούει κανείς να μιλάτε για το θέμα αυτό και ξέρουμε πόσο προσφυλές σας είναι ακόμα και πάντα. Εν τω μεταξύ θέλω να απευθύνω ένα θερμό καλωσόρισμα στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Ταγιάννη. Καλώς ήρθατε σε αυτήν την διάσκεψη και έχουμε κάτι κοινό εδώ, πρόεδρε. Πώς συχνά δεν προεδρεύουμε σε μισοάδιες αίθουσες. Σήμερα βλέπετε την αίθουσα να είναι κατάμεστη. Η κάθε θέση ε, είναι πιασμένη και υπάρχει και κόσμος όρθιος. Ε, αυτό δείχνει πόσο κόσμο έχει ενδιαφερθεί, ότι όλοι γνώριζαν για τη διοργάνωση αυτή τη διάσκεψη και έχουν έρθει εδώ για να ακούσουν για το θέμα αυτό. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είστε εξαιρετικό πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Φίλοι μου, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, ε, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί υποστηκλημένοι, σα ευχαριστώ που ήρθατε και για τη συμμετοχή σα σε, αυτήν τόσο αυτή τόσο σημαντική εκδήλωση. Για το μέλλον τη προάσπιση τη δημοκρατία στον κόσμο. Για μα, η Ευρώπη πάνω απ' όλα σημαίνει ελευθερία, δημοκρατία, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Όχι μόνο Κεντρική Τράπεζα, Ευρώ, Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ευρώπη πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τις αξίες μας και θέλουμε να τις ενισχύσουμε αυτές παντού στον πλανήτη. Θέλουμε να συνεργαστούμε με όλους για την άμυνα αυτή υπέρ της δημοκρατίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποδείξουμε αυτή μα την αφοσίωση σε αυτόν τον σκοπό που στον έχουμε συνταγμένη για την παρατήρηση εκλογών παντού. Και τώρα επιτρέψτε μου να μιλήσω τελικά. Το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει έναν ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό στην παρατήρηση των εκλογών σε όλο τον κόσμο και για να συμβάλλει στην πράσπιση, όπως είπα, της δημοκρατίας. Σε όλες τις χώρες όπου θα μπορούσαν να, υπάρξουν απειλές κατά της λαϊκής βούλησης. Η πρώτη αποστολή έγινε το 1994 στην Λευκορωσία και μέχρι σήμερα είχαμε 209 αποστολές παρατήρησης εκλογών από το Κοινοβούλιο σε 78 χώρες. Οι αποστολές αυτές είναι και ένα παράδειγμα της απόλυτης αφοσίωσής μας στην ε, εύρωστη κοινοβουλευτική διπλωματία, ένα εργαλείο ζωτική σημασίας για να μπορέσουμε να έχουμε και μια σημαντική παρουσία στο διεθνές προσκήνιο πάντοτε ε, με μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ε, προσήλωση κοιτάζουμε πώς οι βουλευτές όχι μόνο της δικής μας της Ένωσης αλλά όλου του κόσμου ε, γιατί εκεί βρίσκεται η εξουσία του λαού συμπεριφέρονται. Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι των εθνών, όχι μόνο οι κυβερνήσεις αλλά οι βουλές, τα κοινοβούλια όπου εκατοντάδες γυναίκες και άνδρες εκπροσωπούν τους πολίτες. Και βεβαίω ε, είναι προ όφελο των πολιτών μα να έχουμε κόσμο με περισσότερη δημοκρατία και λιγότερα από τα αρχικά καθεστώτα. Ε, σταθερότητα, και το βλέπουμε αυτό με του μετανάστε, την οικονομική κρίση, δείτε τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα ή σε τόσα άλλα μέρη του κόσμου. Το να παρακολουθούμε τι εκλογέ σε τρίτε χώρε απαιτεί αξιοπιστία και πολιτική ευαισθησία. Στην Λιβύη μα το ρώτησαν εγώ την επισκέφθηκα τη χώρα, χώρα με πολλές δυσκολίες, με μεγάλα προβλήματα και πολλή αστάθεια. Ε, μου το ζήτησαν να στείλω ευρωβουλευτέ για να παρατηρήσουν τις εκλογές στην επόμενη διοργάνωσή τους. Το γεγονός ότι η δράση αυτή έχει οργανωθεί από εκπροσώπους εκλεγμένους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει μεγάλη προστιθέμενη αξία στην όλη, ε, στην όλη διοργάνωση της παρατήρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν στις αποστολές της έχει πάντοτε έναν επικεφαλής παρατηρητή και ε, αυτός είναι πάντα ευρωβουλευτής ε, σε θέση να αξιολογήσει τις ε, τεχνικές πληροφορίες και να διεξαγάγει τα ανάλογα πολιτικά συμπερόσματα. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι το μόνο διεθνής οργανισμός που παρατηρεί εκλογές σε τον κόσμο μαζί με τον ΟΑΣΕ αλλά και με την Υπηρεσία για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα, δικαιώματα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον ΟΔΙΡ, στον υπόλοιπο κόσμο με την ε, σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λόγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάσκεψη σήμερα έχει σκοπό να βοηθήσει το Ευρωκοινοβούλιο να αναλάβει όλες αυτές τις υποχρεώσεις με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να παίξει ένα ρόλο πιο καθοριστικό στην προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Δυσκολίες που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολλέ ε, μεταξύ άλλων και λόγω των νέων τεχνολογικών μέσων και των νέων μέσων επικοινωνία. Η Μαρία Γκάμπριελ μας παρουσίασε τις ευκαιρίε, αλλά και του κινδύνου που έχουν να κάνουν ε, με τον ψηφιακό κόσμο. Θέλω να την ευχαριστήσω για την δουλειά που κάνει για την ε, προάσπιση της δημοκρατίας και Τη ελευθερίας της χώρας μας, για την καταπολέμηση των ε, ψευδών ειδήσεων σε πολλές χώρες του κόσμου και στην Ευρώπη. Πρέπει να αναχαιτήσουμε την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο ε, και ιδίως σε προεκλογικές περιόδους. Είναι πραγματικά σημαντικότατο αυτό. Έχουμε την ανάγκη να ακούσουμε όλους εδώ και νομίζω ότι ο κύριος ε, Μακάλιστερ είναι ο καλύτερος ε, εκφραστής του Κοινοβουλίου μας για να μπορέσει να, να συγκεφαλαιώσει όλες τις παρατηρήσεις, τα αιτήματα, τις ιδέες και τις επτά επικριτικά σχόλια και αυτά είναι ευπρόσδεκτα μπορούν να μα βοηθήσουν να βελτιωθούμε. Γιατί θέλουμε να προσφέρουμε στη διεθνή κοινότητα, να βρούμε έναν τρόπο να αποστείλουμε μηνύματα φιλίας στι υπόλοιπε χώρε του κόσμου και να δώσουμε και κάτι. Αλλά αν κάτι δεν πάει καλά, αν κάτι πρέπει να το διορθώσουμε, να το βελτιώσουμε, να το κάνουμε. Ε, πάντοτε είμαστε πρόθυμοι να ακούμε και επικριτικά σχόλια, παρατηρήσει ιδέε για να βελτιώσουμε τη δουλειά μα. Είναι τόσοι οι βουλευτέ που έχουν σωρεύσει πλέον μακρά πείρα ε, ως ε, παρατηρητές εκλογών. Και αυτό είναι σημαντικό να μας πείτε και εσείς πώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο είμαστε οργανωμένοι και ε, έχουμε διατάξει τις εργασίες μας. και στις πρεσβείες των χωρών που ενδιαφέρονται, που διεξάγονται εκλογέ, εκεί οι εκπρόσωποι μας είναι διαθέσιμοι για να υπάρξει μια αγαστή συνεργασία. Εύχομαι λοιπόν να εργαστούμε καλά και να ε, καλλιεργήσουμε αυτήν την ε, σχέση, την αμφίδρομη σχέση. Σας ευχαριστώ λοιπόν που βρίσκεστε εδώ, ευχαριστώ όλους τους προκεκλημένους μας, ευχαριστώ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και όλους μας τους βουλευτές που έχουν αναλάβει δράση σε αυτόν τον χώρο και η διάσκεψη αυτή δεν θα είναι απλώς ε, μια επίσημη διάσκεψη ανώτερου επίπεδου, αλλά θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε και την ποιότητα των επόμενων αποστολών μας για την παρατήρηση εκλογών. Αυτό προ όφελο της Ευρώπης της ίδιας, προ όφελο των χωρών που θα μας υποδεχτούν, αλλά πάνω απ' όλα προ όφελο της προάσπισης και της άμυνας της δημοκρατίας και της ελευθερία και της λαϊκή βούληση ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι που κι εσείς ε, εκτιμάτε την εργασία που κάνουμε στον τομέα παρατήρησης των εκλογών και θα βασιστούμε στη βοήθειά σας και για τις επόμενες ε, ε, αποστολές παρατηρήσεων. Ξέρουμε πόσο πολύ άσχολος είστε και θα δώσω τώρα το λόγο στον Αντώνιο Παντζέρη τον συνάδελφό μου που θα παρουσιάσω τους δύο επόμενους ομιλητέ και κατόπιν θα ολοκληρώσουμε, ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ε, περιστοιχίζουμε από ιταλού σήμερα το πρωί. Το απόγευμα, συγγνώμη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ τον πρόεδρο Ταγιάννη που κατάφερε να έρθει. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή μας, θέλω να κάνω και εγώ δύο πολύ ειδικές παρατηρήσεις. Πρώτον, Μπορώ να πω, πιστεύω, ότι η παρατήρηση των εκλογών είναι αναμφίβολα ένα καθοριστική σημασία εργαλείο και δεν είναι και απομονωμένο στο παρελθόν, την τελευταία δεκαετία, ε, ιδίως εμείς οι παρατηρητές, είδαμε να εντείνεται η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση όλων για το ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στην ημέρα μόνο των εκλογών για την εκλογική παρατήρηση, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη ολόκληρο τον κύκλο της προεκλογικής περίοδου ε, για το στόχο αυτό. Όλοι οι διαθέσιμοι πόροι και τα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται για να βεβαιωθούμε ότι η προετοιμασία τη διεξαγωγή των εκλογών είναι άριστη ε, προ όφελο όλων των ε, εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων. Μιλάω τώρα για, την, ε, για τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την διοργάνωση των εκλογών, για τους συμμετέχοντες, τους υποψηφίους, τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους, πολιτικούς, τους τοπικούς Αυτό θα πρέπει να ξεκινά πολύ πριν τι εκλογέ. Και κατά τη διάρκεια τη διαδικασία των εκλογών πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι η δουλειά που έχει γίνει από τι προηγούμενες ε, αποστόλες παρατήρηση, οι μελέτες, οι συστάσει ε, τηρούνται και εφαρμόζονται προκειμένου να βελτιώσουμε την διεξαγωγή των ε, μελλοντικών εκλογών και έτσι να ενισχυθεί η δημοκρατία, η που βασίζεται στι εκλογέ. Αλλιώ ε, γινόμαστε σαν το σύσυφο και προσπαθούμε να σπρώχνουμε την ίδια πέτρα ε, ξανά και ξανά στον ανήφορο. Το Ευρωκοινοβούλιο με τη δουλειά του για την υποστήριξη της δημοκρατίας και τον συντονισμό ε, των εκλογών ε, ομάδα όπου θα σας έχει αναφέρει και ο πρόεδρος Μακάλιστερ στις παρατηρήσεις του έχει ξεκινήσει να προσπαθεί να κάνει αυτή τη δουλειά ε, διοργάνωσης με όσο το δυνατόν ε, πιο συντονισμένο τρόπο και για να έχουμε βιώσιμα αποτελέσματα στις διάφορες προσπάθειες στήριξης της δημοκρατίας και παρατηρήσεων του εκλογικού κύκλου. Αυτό συμπεριλαμβάνει βεβαίω και την παρατήρηση των εκλογών και την ε, συνέχεια που δίνεται στην τήρηση των συστάσεων των παρατηρήσεων που ήδη έχουν γίνει, τι διαδικασίε οικοδόμηση δυνατοτήτων, την πρόληψη συγκρούσεων, τι δράσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δουλειά με τα πολιτικά κόμματα και με νέους πολιτικούς ηγέτες και τι ε, δράσει διαμεσολάβηση, διευκόλυνση και διαλόγου, τι πρωτοβουλίε διαλόγου στις διάφορες χώρες. Έπειτα στην Υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα επικεντρωνόμαστε και στον αντίκτυπο του εργαλείου για την παρατήρηση, την παρατήρηση εκλογών, στις χώρες όπου αυτές διεξάγονται για να είμαστε αποτελεσματικοί, εκλογική παρατήρηση πρέπει να γίνεται αντιληπτή και από τη χώρα υποδοχής ως ένα εργαλείο δημοκρατίας, μάλιστα μακρόπνο, μακροπρόθεσμο, για να, που θα έχει σκοπό να προσφέρει θετικές αλλαγές και να προτείνει μεταρρυθμίσεις εκεί που υπάρχουν ε, κενά στο δημοκρατικό σύστημα της τρίτης χώρας και πάνω απ' όλα να βοηθήσει να καλλιεργηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών αυτό για μας στην Ευρώπη είναι προτεραιότητα. Κατά τη διάρκεια των ε, παρατηρήσεων λοιπόν εκλογών θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας αυτό το σημείο. Το δεύτερο θέμα που θέλω να σας αναπτύξω πριν δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας είναι ότι είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να κατανοούν ότι το εργαλείο παρατηρήσεων εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πραγματικά ένα διαθεσμικό εργαλείο ένα εργαλείο στο οποίο συμμετέχουν όλα τα βασικά θεσμικά όργανα της Ένωσης κάθε απόφαση να αποσταλεί ε, αποστολή παρατήρησης εκλογών τη Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε διαβουλεύσεις και ε, συνεννοήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου. Κάθε αποστολή παρατήρησης εκλογών ε, είναι υπό την ε, ευθύνη ενός μέλους του Ευρωκοινοβουλίου που είναι ο επικεφαλής παρατηρητής και τον οποίο διορίζει αντιπρόεδρος ή πατεκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ε, συνέχεια που δίνεται στις αποστολές είναι κάτι που φροντίζουν οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, στην οικία χώρα ε, με, την τον ανάλογο πολιτικό διάλογο και τα εργαλεία συνεργασίας που έχουμε. Στη, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενημερωνόμαστε μεταξύ μας για τις σχετικές δράσεις παρατήρησης εκλογών και τις καλλιεργούμε, τις ε, αναπτύσσουμε μαζί. Πιστεύω ότι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του εργαλείου για την παρατήρηση εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς αυτή η στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ε, και η Αφρικανική Ένωση αποστέλει αποστολές παρατήρησης εκλογών, θα ήταν καλό να ακούσουμε και τις δικές σας εμπειρίες, το τι έχετε συναντήσει επιτόπου στην πράξη. Έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία ε, Σεσούμα Μινάτα Σαμάτε, επίτροπο για τις πολιτικές υποθέσεις της ε, Αφρικανικής Ένωσης, η οποία είναι δικηγόρος και διπλωμάτης και έχει υπάρξει διευθύντρια στον μηχανισμό, τον μεικτό μηχανισμό συντονισμού και στήριξη τη υβριδική αποστολή τη Αφρικανική Ένωση και του ΟΗΕ για τον Ταρφούρ. Υπήρξε πρέσβυρα στην Μπουργκίνα Φάσο και στην Αιθιοπία, τη Μπουργκίνα Φάσο μάλλον στην Αιθιοπία και μόνιμη εκπρόσωπο τη Αφρικανική Ένωση, καθώ και υπουργό περιφερειακή ανάπτυξη στην Μπουργκίνα Φάσο και ε, σύμβουλο διπλωμάτη του Προέδρου παρά το πρόεδρο στην Μπουρκίνα Φάσο. Σας δίνω το λόγο για τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να χαιρετήσω τον πρώτο κοινοβουλίου που ήδη αποχώρησα και όλα τα μέλη του Προεδρείου. Όταν άκουσα την κυρία Γκάβριελ συμφώνησα με αυτά που είπε για την παρατήρηση των εκλογών. Και εμείς ως Αφρικανική Ένωση πιστεύουμε τα ίδια πράγματα. Πριν όμως σας ενημερώσω για την πείρα της Αφρικανικής Ένωσης, χαιρετίζω όλους τους, ε, τους συμμετέχοντες. Ε, βλέπω διάφορες διακεκριμένες προσωπικότητες που τους έχω συναντήσει και κατά τη διάρκεια αποστολών παρατηρήσεων και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων της Ένωσής μου. Και θέλω να χαιρετήσω λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προσκάλεσε την ε, Αφρικανική Ένωση σε αυτήν την ε, σημαντική εκδήλωση υψηλού επίπεδου για το μέλλον των αποστολών παρατηρήσεως εκλογών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, της Αφρικανικής Ένωσης, ο κύριος Φακή, ήθελε να είναι ο ίδιος παρόν για να σας ενημερώσει αλλά λόγω άλλων ανηλυμένων υποχρέσεων δεν είναι παρόν αλλά εύχεται πλήρη επιτυχία στις ε, συζητήσεις μας. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν φίδεται προσπαθειών για να ενισχύσει την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο οργανώσεών μας. Είμαι χθες, από χθε εδώ, έχω κάνει πολλές επαφές με διάφορους επιτρόπους για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών. Και πολύ συχνά συναντιόμαστε και στις διάφορες αποστολές και ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Κυρίες και κύριοι, στην Αφρική κάθε χρόνο γίνονται 15 με 20 εκλογές. Κοινοβουλευτικές, προεδρικές και θα μπορούσαμε να, είναι, να πούμε ότι είναι και περισσότερες γιατί έχουμε και αυτοκι, αυτοδιοικητικές εκλογές καθώς και δημοψηφίσματα όπου δεν αποστέλουμε παρατηρητές. Εκτός εάν πρόκειται για το νότιο Σουδάν όταν το ερώτημα ήταν αν θα γίνει ανεξάρτητο κράτος. Τότε ήμασταν παρόντες. 15 με 20 εκλογές το χρόνο αυτό αποδεικνύει πόσο οι Αφρικανοί εκτιμούν τις ε, δημοκρατικές αρχές. Και βέβαια θα θυμάστε ότι κάποια άλλη στιγμή ε, αντί γι' αυτό γίνονταν πολλά δημο, ε, συγγνώμη, ή κυβερνητικές αλλαγές αντιδημοκρατικές. Έχουμε μία μοναδική χάρτα, μία χάρτα για τη δημοκρατία και τις εκλογές. Και αυτή η χάρτα είναι η βάση μας για τη λειτουργία όλων των αποστολών παρατήρησης στην Ήπειρό μας. Τι έγινε το 18. Η Επιτροπή μας παρακολούθησε γύρω στις 20 εκλογές, συγκεκριμένα 19. Αλλά επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμη ο χρόνος, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπερβούμε τις 20 και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να το κάνουμε. Οι περισσότερες εκλογές λοιπόν που θα παρατηρήσουμε φέτος έχουν ήδη λάβει χώρα και στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό επικίνδε. Και του χρόνου θα έχουμε πολύ σημαντικές εκλογές, όπως για παράδειγμα στην Ιγυρία, την Νότια Αφρική. Και φυσικά θα είμαστε παρόντες ως ε, Αφρικανική Ένωση ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την πρόοδο της δημοκρατίας στην Ήπειρό μας. Στο παρελθόν οι αποστολές αυτές ήταν πολύ τεχνικές, αλλά επειδή υπήρχαν πολλές αμφισβητήσεις για τις αποστολές αυτές, δώσαμε περισσότερο βάρος στην προληπτική διπλωματία. Ήδη αναφέρθηκε αυτό το θέμα. Εξετάζουμε κάθε φάση της εκλογικής διαδικασίας και δημοσιοποιούμε τα πορίσματά μας. Είμαστε παρόντες πριν, κατά και μετά. Αλλά παρακολουθούμε και τι γίνεται εκ των υστέρων. Γιατί μετά από ορισμένε εκλογές ε, πολλές φορές προκύπτουν ε, κρίσεις. Πολλές φορές οι κρίσεις στην Ήπειρό μας προκύπτουν από εκλογές. Το μέλλον της διεθνούς παρατήρησης εκλογών απαιτεί από όλους μας μία αυξημένη δέσμευση από τα κράτη-μέλη και μία βελτίωση των μεθόδων μας. Και ε, θα ήθελα να παίξει μεγαλύτερο ρόλο η προληπτική διπλωματία. Το υπογραμμίσατε κι εσείς κυρία Γκάμπριελ, χρειάζεται συνεργασία μεταξύ θεσμών, αλλά και μεταξύ των περιφερειακών οικονομικών κοινοτήτων που έχουμε στην Αφρική. Αυτό πρέπει να γίνει απαραίτητο, γιατί οι κρίσει μας, σας είπα πολλές φορές, προκύπτουν από όχι καλά διεξαρθήσει εκλογές. Και υπάρχουν και συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί. Στις 17 Απριλίου 2017 υπογράψαμε μια συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη για την κυβερνοασφάλεια και τη διακυβέρνηση. Επίσης, υπογράψαμε μια συμφωνία τον Μάιο του 2018 με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση αυτέ τι δύο συμφωνίε. Έχουμε πλατφόρμες συνεργασίας για να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας, την κοινή μας δέσμευση, για να αποφευχθούν οι κρίσεις που μπορεί να προκύψουν από κακώς διεξαχθήσεις εκλογές, όπως είπα και προηγουμένως. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια οι οργανώσεις μας και χαιρετίζω και την ε, αδελφοί μου από την ε, Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συνεργαστεί. Την τελευταία φορά που τα πήγε πολύ καλά αυτή η συνεργασία ήταν στη Ρουάντα. σα ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και στο Ζιμπάμπουε μαζί επίσης συνεργαστήκαμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκύψουν κρίσεις. Βεβαίω, ε, ο συνδυασμό προσπαθειών δεν σημαίνει και απώλεια αυτονομίας. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, δεν χάνουμε το χαρακτήρα μας, την ανεξαρτησία μας. Ούτε χάνουμε το δικαίωμα να πούμε την αλήθεια για αυτά που παρατηρήσαμε επί τόπου όπου διεξάγονται εκλογές. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών. Και πριν και μετά, ούτως ώστε να διαμορφώνουμε κοινέ στρατηγικές που να μας επιτρέπουν να αποφεύγουμε λοιπόν τις κρίσεις στα αφρικανικά κράτη μετά τις εκλογές. Επίσης, θεωρούμε ειλικρινά και νομίζω ότι και εσείς το είπατε, οι αποστολές αυτές σε τι πρέπει να καταλήξουν, σε συστάσεις. Το χαιρετίζω αυτό. Στο μέλλον θα έπρεπε να δούμε πώς θα εφαρμόζονται αυτές οι συστάσεις για να διορθωθούν όσα δεν πάνε καλά. Να μπορέσουν οι ίδιες οι χώρες να τα διορθώσουν με βάση τις παρατηρήσεις μας, με βάση αυτό που είπαμε ότι δεν λειτουργεί σωστά. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη συνεργασία και με τις περιφερειακές οικονομικές κοινότητες όπως είπα που παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Στην περίπτωση της ΣΕΝΤΕΑΟ παίζει τεράστιο ρόλο και η Σαντέκ και η Λίγα και όλες οι άλλες. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με όλες αυτές τις ε, περιφερειακές κοινότητες. Πρέπει να δούμε όμως και την ε, μεθοδολογία μας, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε την παρουσία επαρκών και αποτελεσματικών παρατηρητών σε όλες τις φάσεις της ε, εκλογικής διαδικασίας. Αναφέρεται η τεχνολογία. Βεβαίως η τεχνολογία μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μας δημιουργήσει νέα προβλήματα. Γιατί υπάρχουν ε, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Διότι, όπως ξέρετε, στην Αφρική οι περισσότεροι ψηφοφόροι δεν γνωρίζουν αυτές τις τεχνολογίες. Να πείτε σε έναν ε, ψηφοφόρο που κατοικεί χίλια χιλιόμετρα από την κυβέρνηση να ψηφίσει ηλεκτρονικά, τι σημαίνει. Δεν έχει δει υπολογιστή, δεν γνωρίζει τι είναι, δεν υπάρχει ηλεκτρισμός πολλές φορές. Πρέπει λοιπόν η τεχνολογία να προσαρμόζεται στις ηθίκες της χώρας. Φυσικά πρέπει να ανθαρρύνουμε τη χρήση τεχνολογιών, αλλά να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είδατε τι έγινε στην Κένια. Υπήρξαν δυσχέρειες. Βεβαίως εθαρρύνουμε τις τεχνολογίες, αλλά να βασιστούμε στη σωστή τεχνογνωσία για να μπορούμε να εκτιμούμε πώς έχει η κατάσταση επιτόπου. Να αξιολογήσουμε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την χρήση των νέων τεχνολογιών. Ε, πολλοί αναφέρθηκαν και στο ρόλο των μέσων. Παίζουν ρόλο επιτόπου. Βεβαίω οι ψευδείς ειδήσει παίζουν το ρόλο τους. Γιατί μπορεί να παίξουν αρνητικό ρόλο στην εκλογική διαδικασία. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Εμείς ως Αφρικανική Ένωση αποστέλουμε και μακροπρόθεσμες και βράχοι πρόθεσμες αποστολές και αποστολές παρακολούθησης για το τι θα συμβεί μετά και αποστολές υψηλού επίπεδου. Στι αποστολέ υψηλού επίπεδου συνήθω επικεφαλή είναι ένας πρώην πρόεδρο Αφρικανική χώρα ή ένα ε, ε υπουργό, ε, μια προσωπικότητα εξέχουσα. Και χαιρετίζω και τον πρόεδρο του ΠΑΠ που είναι εδώ παρόν. Έχουμε και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που συμμετέχει. Είναι δηλαδή αποστολές όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι πολλών οργάνων για να έχει και καλά αποτελέσματα. Και επίσης, όλο και περισσότερες είναι αυτές οι αποστολές υψηλού επίπεδου. Επικεφαλής είναι ο πρόεδρος Φακή και αν δεν είναι διαθέσιμος τότε πηγαίνω εγώ επικεφαλή, πολλές φορές πάμε μέχρι και 20 για να διασφαλίσουμε να γίνουν σωστά οι εκλογές και να γίνουν αποδεκτά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και αν δεν γίνονται αποδεκτά, να μπορέσουν να, γίνουν, ε, να υπάρξουν ε, δικαστικές διαδικασίες αμφισβήτηση και όχι διαδηλώσει στους δρόμους για να μην έχουμε νεκρού. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με όλους τους φορείς στην Ήπειρό μας και αυτή η συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω συνεργασίας με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση για την βοήθεια που έχει δώσει στην Αφρικανική Ένωση. Γιατί, όπως ξέρετε, το 2013 ξεκινήσαμε την προσπάθεια εκπόνησης ε, μεθοδολογίας ε, μακροπρόθεσμης διάρκειας ούτως ώστε να αποφεύγουμε τις ε, συγκρούσεις εντοπίζοντας τις δυσχέρειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις. Και έτσι έχουμε αποκτήσει περισσότερη αξιοπιστία και εμείς και οι εκλογικές διαδικασίες αυτές. Και θέλουμε οι εκθέσεις τις οποίες δημοσιεύουμε να περιέχουν όλα τα ουσιώδη στοιχεία. Δεν είναι κανένα θέμα ταμπού. Έχει τελειώσει η περίοδος όπου βλέπαμε διάφορα περίεργα πράγματα και δεν τα βάζαμε σε εκθέσεις μας. Τώρα είμαστε πεπισμένοι ότι οι δημοκρατικές αξίες πρέπει να αναφέρονται και να τηρούνται αυτά που είπαμε. Γιατί ε, είχαν επικριθεί οι αποστολές ότι έκαναν συστάσεις που δεν είναι ρεαλιστικές. Και εγώ συμφωνώ. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι ρεαλιστικές, που δεν εφαρμόζονται. Το βασικό λοιπόν είναι οι αποστολές αυτές να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο από την Αφρικανική Ένωση για να αποφύγουμε κακές εξελίξεις. Για παράδειγμα στο Μαλί έγιναν εκλογές και σήμερα η κατάσταση είναι δύσκολη. Στο Καμερούν ε, είναι εν εξελίξει διαδικασία και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. στο Μαλί που ήμουν παρούσα, μετά φύγαμε. Όχι, έπρεπε να παραμείνουμε εκεί για να βοηθήσουμε τον κόσμο εκεί να αποφύγει τα χειρότερα. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στην παρουσία μας. Και δεν αμφιβάλλω, κυρίες και κύριοι, ότι η διεθνής παρατήρηση των εκλογών θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της, όπως γίνεται και τώρα, αλλά πολύ περισσότερο στο μέλλον. Και για να έχουμε αξιοπιστία, Πρέπει να εξελιχθούμε, να είμαστε δημιουργικοί. Αν δεν τα κάνουμε αυτά, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Και οι περιφερειακοί θεσμοί και οι διεθνείς οργανισμοί όλοι πρέπει να είμαστε απαραίτητοι. Και κυρίως πρέπει να αυξήσουμε την αξιοπιστία των εκλογικών διαδικασιών και την αποδοχή από όλους των αποτελεσμάτων. Παντού και ιδιαίτερα στην Αφρική. Αυτά για να σας εξηγήσω τι κάνουμε ως Αφρικανική Ένωση και όταν ακούω αυτά που κάνετε ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κοινέ αξίες, καταλήγουμε στα ίδια πορίσματα και θα συνεχίσουμε από κοινού, θεωρώ, τον αγώνα για την ε, ανάπτυξη της δημοκρατίας, της αναδυόμενης ε, δημοκρατίας στην Υπηρώμα. Ε, μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία Σαμάτε για την ε, ομιλία σας. Τώρα, τελευταίος ε, για την εναρκτήρια αυτή μας Πάση τη συνεδρίαση, η κυρία Σάλε Βέντε, υπογραμματέα, ε, γενική γραμματέας και ειδική επεσταλμένη στην Αφρικανική Ένωση του ΟΗΕ, επίσης επικεφαλής της υπηρεσία για την Αφρικανική Ένωση του ΟΗΕ και υπήρξε υπεύθυνη του Γενικού Γραφείου της Γενικής Υπηρεσία του ΟΗΕ στο Ναϊρόμπι, ειδική εκπρόσωπο και επικεφαλή του ΟΗΕ για τις Επιρεσίες διατήρηση της Ειρηνή. Ε, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και μόνιμη εκπρόσωπο της Αιθιοπίας στην Αφρικανική Ένωση, καθώς και μέλο τη ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για την Αφρική του ΙΕ. Επίση, Γενική Διευθυντή ε, για τι Αφρικανικέ Υποθέσει ε, στο Υπουργείο Εξωτερικών τη Αιθιοπία, πρέσβυρα τη Αιθιοπία στην Γαλλία και μόνιμη εκπρόσωπο στην UNESCO. Γι' αυτό σας, θα σα ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να χαιρετήσω την επίσημη παρουσία της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Προεδρείο. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση που απίφθηνε στην Ηνωμένα Έθνη να ε, μιλήσουμε σε αυτό το εκλεκτό ακροατήριο σήμερα. Με χαρά βρίσκομαι εδώ. Ποιος είναι ο στόχος της διάσκεψης. Είναι και κρίσιμος και επίκαιρος. Πριν συζητήσουμε για το μέλλον, επιτρέψτε μου σύντομα να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν. Πριν από 13 χρόνια, το Οκτώβριο του 2005, υπήρξε η ε, αρχή διακήρυξη, η διακήρυξη στα Ηνωμένα Έθνη, στα έδρα του ΟΗΕ, για την παρατήρηση εκλογών. Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας ε, να αποτελέσει αυτό ένα δεσμευτικό μέσο των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μάλλον ένα σύνολο κατευθυντήριο ε, γραμμών που από κοινού και με λογική έχουμε εκπονήσει για να αυξηθεί η συνέπεια, η αμεροληψία και ο επαγγελματισμός κατά τη διάρκεια της παρατήρησης εκλογών. Για να γνωρίζουμε και ποια είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των διεθνών παρατηρητών. Μεταξύ άλλων αυτά περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για υψηλά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς, αρχές αμεροληψίας και σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, αλλά και ανεξαρτησία και ευθύνη στην αξιολόγηση των ευρημάτων καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής ε, αναμέτρησης. Και όλα αυτά να αποτελέσουν τη βάση για επικοδομητικές συστάσεις έτσι ώστε να βελτιώνονται οι μελλοντικές εκλογές. Οι αρχές αυτού του κώδικα δεοντολογίας εμπνέονται από μία αίσθηση ε, κοινή ευθύνη. Ο τότε πρόεδρος ε, Κόφι Ανάν ανακοίνωσε τον κώδικα συμπεριφοράς και τόνισε ότι η αποστολή παρατήρησης εκλογών είναι πάντα μετά από ε, πρόσκληση των αρχών της εκάστοτε χώρας και μπορεί να βοηθήσουν στον εκδημοκρατισμό ε, της χώρας και μόνο η παρουσία τους ε, εμπνέει εμπιστοσύνη γιατί αποτρέπει ε, τις δυσλειτουργίες της εκλογικής διαδικασίας. Αυτό συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη. Το πνεύμα ποιο είναι, ότι οι παρατηρητές των εκλογών πάντα συνεισφέρουν θετικά. Αυτό όλο ήταν παράθεση της ομιλίας του Κόφιαναν. Η εκλογική υποστήριξη στα κράτη-μέλη το Ηνωμένων Εθνών ήταν πάντα σημαντικό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ε, λήξης απεικιοκρατίας ε, και της ανεξαρτησίας πολλών κρατών παρατηρήσαμε τα δημοψηφίσματα που οδήγησαν ε, στη δημιουργία νέων κρατών. Σήμερα οι αποστολές παρατήρησης εκλογών σπανίως χρειάζονται εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας ή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μάλλον τεχνική βοήθεια ε, παρέχουμε στα κράτη-μέλη, 60 το αριθμό αυτή τη στιγμή. Όταν μας ζητούν τις καλές μας υπηρεσίες για την υποστήριξη αξιόπιστων διαδικασιών και ειρηνικών εκβάσεων. Ο σημαντικός ρόλος των διεθνών παρατηρητών εκλογών για την αύξηση ε, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της δημόσιας εμπιστοσύνης στις εκλογικές αναμετρήσεις ε, τώρα είναι κάτι που έχουν απομειστεί σε μεγάλο βαθμό περιφερειακοί οργανισμοί. Στη τελευταία έκθεση, ο Γενικός Γραμματέας ε, ανέφερε στη Γενική Συνέλευση με ικανοποίηση ότι όλο και περισσότερα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τις εκλογές ως ειρηνικό μέσο έκφρασης της λαϊκής βούλησης. Ταυτόχρονα όμως σημείωσε την αυξανόμενη περιπλοκότητα και τις προκλήσεις. Οι εκλογές σε κάποιες σπάνιες πλην τραγικές περιπτώσεις ε, αντί να φέρουν την ειρήνη πυροδοτούν ένοπλες σειράξεις. Υπάρχουν ε, κάποιοι που εκμεταλλεύονται τις εκλογές για να επιτύχουν τις πολιτικές τους επιδιώξεις. Ε, και αρνούνται τα αποτελέσματα των εκλογών που εκφράζουν λαϊκή βούληση. Στις νέες τεχνολογίες και τα social media με την ε, αυξημένη χρήση τους ε, μπορεί να έχουμε ευκαιρίες αλλά και κινδύνους που πρέπει εκ των προτέρων να αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να συμμετέχουν με νόημα και οι γυναίκες και οι νέοι, ε, τα άτομα με αναπηρίες και ομάδες που παραδοσιακά είναι περιθωριοποιημένες. Είναι αυτές οι προκλήσεις και άλλες ε, βέβαια είναι στα χέρια των κυρίαρχων ε, κρατών μελών. Όταν μας ζητούν την υποστήριξή μας όμως θα πρέπει να εξακολουθούμε να εκτελούμε τα καθήκοντά μας με σεβασμό, με συνέπεια, με απεροληψία και με τα ε, ύψιστα πάντα επαγγελματικά πρότυπα. Υπό το πνεύμα αυτό λοιπόν της συλλογική ευθύνη καταλήξαμε το 2005 στη Νέα Υόρκη ε, στη διακήρυξη αυτή αρχών ε, για την οποία συζητούμε και σήμερα. Ο Γενικός Γραμματέας ε, Αντώνιο Γκουτέρες στη Γενική Συνέλευση ε, μίλησε ε, για το πόσο πεπισμένος είναι για την πολυμερή προσέγγιση σε ένα κόσμο πολύ πολικό σήμερα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις εταιρικές σχέσεις και τη συνεργασία μας και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση. Πρόσφατα συνάψαμε μια συμφωνία για στρατηγική και συνεργασία για ε, ειρηνευτικές ε, αποστολές και διαχείριση κρίσεων και την ε, ατζέντα του 2063 και την ατζέντα για το θεματολόγιο μάλλον για την βιώσιμη ανάπτυξη. Δείχνουν όλα αυτά πόσο προσιλωμένοι είμαστε στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια και συμμετοχή των βουλευτών για την παρατηρήση των εκλογών. Οι πολιτικοί ηγέτες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση φέρουν πάντα την ευθύνη για την επιτυχία των εκλογών. Θα πρέπει οι ηγέτες να δεσμεύονται δημόσια, όπως και οι οπαδοί τους, ότι θα, θα σέβονται τις εκλογές και αν έχουν πρόβλημα με το εκλογικό αποτέλεσμα θα πρέπει να προσφεύγουν μόνο στα ένδικα μέσα που προβλέπονται και να δείχνουν ε, μεγαλοψυχία στη νίκη και σεβασμό σε περίπτωση ήττας. Ποιος μπορεί καλύτερα να συζητήσει αυτά τα θέματα με τους πολιτικούς ηγέτες από εκείνους που έχουν ήδη ζήσει τα σκαμπανεβάσματα της ζωής ως ερετή ε, Όπως ακούστηκε και προηγουμένως, η πρόληψη ε, μιας κρίσης είναι το σημαντικότερο και από τις ύψιστες προτεραιότητες των ΟΕΕ και του Γενικού Γραμματέα και είναι και καθημερινή ε, δουλειά και τμήμα της Γενικής Στρατηγικής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόθεσή τους. Το τμήμα πολιτικών υποθέσεων ε, έχει ακριβώς ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη και υποστηρικτικό προς το Γενικό Γραμματέα και των απεσταλμένων του για την πρόληψη κρίσεων. Τα Ηνωμένα Έθνη επίσης συνεργάζονται στενά με περιφερειακούς και άλλους οργανισμούς ε, στις πρώτες γραμμές ε, της πρόληψης των συγκρούσεων. Τέλος, έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι η ε, διεθνή παρατήρηση εκλογών εκφράζει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας να διεξάγονται δημοκρατικά οι εκλογές ως τμήμα του γενικότερου εκδημοκρατισμού. Όταν οι εκλογές γίνονται ε, αμερόληπτα και υπεύθυνα, η εκλογική παρατήρηση μάλλον, είναι πολύτιμο εργαλείο για να αξιολογούνται οι εκλογές σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές για τις γνήσιες ε, και ελεύθερες εκλογές και το δίκαιο δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι οι εκλογές ανήκουν στους πολίτες των χωρών που υπηρετούμε. Οι εκλογές και η δημοκρατία είναι δική τους υπόθεση. Αλλά ε, όταν μας ζητούν τη βοήθειά μας και όσο μας τη ζητούν θα πρέπει να εξακολουθούμε να κάνουμε το καθήκον μας με σεβασμό, με ευθύνη, με συνέπεια και με αμεροληψία και πάντα με ε, το μεγαλύτερο δυνατό επαγγελματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενή σας προσοχή. Ευχαριστούμε σας. Ευχαριστώ πολύ για την ε, σας. Τώρα πρέπει να κλείσουμε αυτή την φάση της συνεδρίασης, της διάσκεψης. Αλλά προηγουμένως θα κάνω μια μικρή παρατήρηση ήδη συμπεράσματος. Σήμερα ακόμη και να επικεντρωνόμαστε σε ένα μόνο εργαλείο για την ε, παρατήρηση των εκλογών, θα πρέπει να έχουμε υπόψη το εξή. Το συνολικό πλαίσιο εργαλείων με το οποίο έχουμε αυτό το ψηφιδωτό, αυτό το πλωστάσιο εργαλείων και τις ψηφίδες ε, για, το, για την προάσπιση της δημοκρατίας Είναι σημαντικό. Θα σας καλέσω λοιπόν στα επόμενα πάνελ να είστε ανοιχτόμυαλοι, λέει και ε, να μην διστάσετε να πείτε τι πηγαίνει καλά και τι όχι στον, στη δικασία παρατήρησης των εκλογών, που υπάρχουν δυσκολίες και αν είμαστε, και να δούμε ποια, αν έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε τα κακοσκήμενα και να δούμε και που μπορεί να υπάρξει άμεση βελτίωση. Αν μιλάμε για το μέλλον τη παρατήρηση των εκλογών, αυτό το εργαλείο τη πολιτική θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αλλαγή. Γι' αυτό σα παροτρύνω όλου να, να συμμετέχετε στι συζητήσει και με ανοιχτό πνεύμα να μοιραστείτε τι εμπειρίε και τι ιδέε σα. Κλείνει τώρα λοιπόν αυτή η εναρκτήρια φάση και μετά το σύντομο διάλειμμα θα συνεχίσουμε με το πρώτο πάνελ ε, προκλήσεις και ευκαιρίες για την παρατήρηση των εκλογών, ε, πληροφορική, ε, παραπληροφόρηση και χρήση των κοινωνικών μέσων. Καλή συζήτηση για τη συνέχεια. Could I please ask everybody to take their seats so that... Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε την ε, συζήτησή μας. Παρακαλώ καθίστε. Και όποιος θέλει να κάνει συζητήσεις παρακαλώ να βγει έξω. Right. Um, very good. There's no point in me welcoming you here. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας καλωσορίσω, γιατί ήσασταν και προηγουμένως, πριν φτάσω. Χαίρομαι που ε, είσαστε ακόμη εδώ, τώρα που ήρθα. Τώρα, να περάσουμε στις συζητήσεις. Θα έχουμε μια σειρά από συζητήσεις. Στην πρώτη θα προεδρεύσω εγώ. Και εδώ έχω και τέσσερις πολύ έμπειρους συναδέλφους. Θουλουέτα που είναι η κυρία Τάνια Τσουλουέτα που είναι Ιταλίδα που έχει ηγηθεί διαφόρων αποστολών παρατήρηση εκλογών από πλευρά του ο ΑΣΕ, κυρίω στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ασία. Την κυρία Μαρίκτιε Σχάκε, πολύ ενεργό και διακεκριμένο μέλος της φιλελεύθερης ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έχει εργαστεί πολύ και για θέματα δημοκρατίας, εκλογών, έχει ηγηθεί και πέρυσι της ε, αποστολής παρατηρητών στην Κένια παρατηρητό στην Κένια και επίση έχει ασχοληθεί με πολλά ψηφιακά θέματα. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν η παρουσία της επειδή συζητάμε το ρόλο της ε, πληροφορικής στις εκλογικές διαδικασίες. Ο Ιβλιο Τέρμ, πρώην υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τελικά προτίμησε να γίνει Πρωθυπουργό του Βελγίου. Και τώρα είναι επικεφαλής του Διεθνούς Ινστιτούτου IDEA για τη δημοκρατία και τις ε, εκλογές με βάση τη Στοχόλμη. Και τελευταίος, αλλά αξίω σημαντικός, ο κύριος Πατ Μέρλερ, που είναι επικεφαλής ε, εκλογικών προγραμμάτων στο Διεθνές Δημοκρατικό Ινστιτούτο, που θα πρέπει να είναι πρωταλλητής από πλευράς ε, αποστολών παρατηρητών στις οποίες έχει συμμετάσχει και έχει συγγράψει και τις καθευτήρες γραμμές για την παρατήρηση εκλογών. Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ γύρω από αυτό το Προεδρείο. Το θέμα μας λοιπόν είναι τεχνολογία τη πληροφόρηση, αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η χρήση των κοινωνικών μέσων. Υπάρχουν ε, πολλές προκλήσεις αλλά και δυνατότητες που μας δίνει η πληροφορική. Ένα καλό παράδειγμα ήταν οι εκλογές στην Κένια πέρυσι όπου κατέρευσε το ψηφιακό σύστημα και το ανώτατο δικαστήριο ζήτησε να επαναληφθούν οι εκλογές. Και αυτό είχε διάφορες πολιτικές επιπτώσεις. Ε, εντάσεις Μείωση της εμπιστοσύνη του κοινού στην εκλογική διαδικασία. Σοβαρή μείωση. Οπότε θα πρέπει και εμείς να δούμε πολύ προσεκτικά τι επιπτώσεις έχει η ψηφιοποίηση των εκλογών. Βεβαίω, μπορεί να διευκολύνουν τις εκλογέ. από την γραφή στους εκλογικούς καταλόγους, ε, ταυτοποίηση και στην ίδια την πράξη τη ψηφοφορία και στην καταμέτρηση. Αλλά θέτει και πολλές νέες προκλήσεις. Αξιοπιστία. Κίνδυνη παρέμβαση σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας. Τι ακριβώς δηλαδή πρέπει να εξετάσουμε όταν εξετάζουμε την εκλογική διαδικασία και η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, στις αρχές και βεβαίως υπάρχουν και προκλήσεις που δημιουργούνται από τα κοινωνικά μέσα που αξιοποιούνται όλο και περισσότερο στις προεκλογικές και γενικότερα πολιτικές διαδικασίες. Στις πρώτες μέρες που ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι από τα κοινωνικά μέσα, όλοι θεωρούσαμε ότι έτσι θα υπήρχε περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ελευθερία, περισσότερη συζήτηση στις κοινωνίες μας. Αυτό ισχύει. Αλλά υπάρχουν και περισσότερες ε, δυνατότητες ε, επηρεασμού, ακραίων ε, απόψεων που αποκτούν, περισσότερον, αποκτούν περισσότερη πρόσβαση και υπονόμευση τελικά της διαδικασίας έκφρασης άποψης και διαμόρφωσης άποψης. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης για τη διαδικασία και για το πολιτικό και το οποίο των μέσων γύρω από αυτά και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ανακύπτουν τι επίβλεψη και τι κανόνες πρέπει να υιοθετηθούν για να ρυθμίσουμε την κατάσταση χωρίς να είμαστε υπερβολικοί. Κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ε, κατάπνιξη της συζήτησης. Ή να έχουμε φαινόμενα όπου κάποιοι θα έλεγαν ότι αυτό είναι ε, απαράδεκτη παρέμβαση, ενώ άλλοι λένε ότι είναι απλώς ελεύθερη έκφραση. Πολλοί παρόντες εδώ, έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό, με όλα αυτά τα θέματα, οπότε εγώ δεν θα προσθέσω, δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο. Να ακούσω τα σχόλια και από τους ομιλητές και από τους ε, συμμετέχοντες. Είδατε και ένα σύντομο έγγραφο με μερικά γενικά θέματα που έχει διανεμηθεί σε όλους. Ελπίζω να έχουμε μια ζωηρή συζήτηση και γι' αυτό θα πρέπει να είναι σύντομες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Και κυρίως πρέπει να εστιάσουμε στις ερωτήσεις που επιχειρήσαμε να διατυπώσουμε ή που θα προκύψουν από το πρώτο γύρο ομιλιών. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο σε δύο από τους ομιλητές μας για τα εισαγωγικά του σχόλια. και μετά θα δούμε πώς θα πάμε. Να ξεκινήσω με την Μαρίτια. Όπως είπα, ήσασταν επικεφαλής της αποστολής παρατήρησης εκλογών στην Κένια πέρυσι για τις ε, εκλογές. Όπου εν μέρη η ε, ανεπάρκεια του συστήματος πληροφορικής προκάλεσε επανάληψη των εκλογών. Γιατί το αποτέλεσμα την πρώτη φορά ακυρώθηκε από το δικαστικό σώμα. Πείτε μας, εντοπίσατε που ήταν οι αδυναμίες του συστήματος ε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, για παράδειγμα. Ήσασταν επικεφαλής της αποστολής. Είχατε τα κατάλληλα μέσα για να παρακολουθήσετε αυτή την πλευρά. θεωρήσατε ότι υπήρχαν ανεπάρκειες ε, στα μέσα που είχατε στη διάθεσή σας. Τι ρόλο έπαιξαν όλα αυτά στην εξέλιξη της προεκλογικής εκστρατείας και στη δική σας ε, παρουσία. Α. Θα ήθελα να ρωτήσω για την Τάνια, αλλά έχει φύγει. Ναι. Θαυμάσαι. Ευχαριστώ πολύ, Κρίστια. Είναι πραγματική η χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας καλωσορίζω, γιατί εδώ είναι και το γραφείο μου ε, και η δουλειά μου και να σας μιλήσω για τη δημοκρατία και την... το πόσο επηρεάζει η τεχνολογία το κράτος δικαίου. Είναι προφανώς παγκόσμια η πρόκληση και ενώ εμείς ε, εστιάζουμε σήμερα στις επιπτώσεις της τεχνολογίας τη δημοκρατία ή τις εκλογικές αναμετρήσεις, έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι εγώ βέβαια δανείζομαι την εμπειρία μου από την Κένια, αλλά ε, στην Ευρώπη δεν το έχουμε λύσει και θα πρέπει οπωσδήποτε να βιαστούμε να το λύσουμε. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα λοιπόν από την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων είναι ο κίνδυνος δημιουργίας μαύρων κουτιών ε, με αλγορίθμους, με τράπεζες δεδομένων, όπου κάποιοι διαχειρίζονται ε, κάποια δεδομένα χωρίς κανείς ανεξάρτητος ε, να επιβλέπει όλα αυτά, να τα εποπτεύει ή να υπάρχει λογοδοσία. Ρώτησες, Κρίστιαν, ε, αν κατέρευσε το σύστημα πληροφορική στην Κένια και γιατί. Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε είναι πώς μπορούν κάποιοι μηχανισμοί δημόσιας λογοδοσίας ιδιωτικών εταιριών να είναι αναπόσπαστο τμήμα μιας τέτοιας διαδικασίας ε, εκλογικής. Αναγνωρίσανε ε, αυτή την αδυναμία, γιατί το ανώτατο δικαστήριο της ε, Κένιας δεν κατάφερε να επιβάλει την πρόσβαση στο κεντρικό σερβερ έτσι ώστε να διαπιστωθεί η σωστή διαχείριση των δεδομένων. Εξού και κατέληξε στην απόφαση να επαναληφθούν οι προεδρικές εκλογές. Όταν προσπαθούμε λοιπόν να αντλήσουμε τα διδάγματα από την εμπειρία αυτή στην Κένια για άλλες αποστολές παρατήρηση εκλογών, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι και ο χρόνος έχει τη σημασία του. Δηλαδή, η φάση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Εάν στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στο μνημόνιο συνεννόησης δεν ορίζεις ακριβώς με ποιον τρόπο θα γίνει η δημόσια εποπτεία και πώς θα λογοδοτούν δημόσια ε, οι ιδιωτικές εταιρείες πριν τους ανατεθεί το έργο, τότε πολύ πιο δύσκολα μπορείς αργότερα να το επιβάλλεις. Εκτός από το επιπλέον κόστος, το οικονομικό, μπορεί να υπάρχουν και διενέξεις στα δικαστήρια και να είναι εις βάρος των ε, ψηφοφόρων. Μιλήσατε λοιπόν για την κατάρρευση της τεχνολογίας και ρωτήσατε γιατί έγιναν. Ε, υπήρξαν πολλά επικίνδυνα στοιχεία. Ζητήσαμε ε, να γίνει ένα συνολικός έλεγχος, μια δοκιμή της τεχνολογίας πριν χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν διάφορα προφανή πράγματα όταν ε, αναπτύσσεις νέα συστήματα ε, σε περιοχές που δεν είναι μεγάλη η κάλυψη σε διαδικτύου ή τηλεπικοινωνίε λειτουργούν σωστά. Όλα αυτά χρειάζονται και θα πρέπει και ο κόσμο να εκπαιδεύεται για να λυθούν τα προβλήματα και όχι τη μέρα των εκλογών αλλά προηγουμένω. Πολύ σημαντικό. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Τα δεδομένα αυτά που διαχειρίζονται οι ιδιοκτήτες του συστήματος ε, πρέπει να ξέρουμε πώς γίνεται αυτή η διαχείριση, ποιος έχει πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους, στα δεδομένα των ψηφοφόρων και να γίνονται όλα αυτά σύνομα. Στην Κένια ε, δεν υπάρχουν νόμοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και όταν τέτοιοι νόμοι δεν υπάρχουν, που συνήθως δίνουν ασφαλιστικές δικλείδες για τα πρόσωπα και υπάρχουν απαιτήσει για το πώς χειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα, λείπουν πλήρως στην Κένια όλα αυτά. Και μία από τις ε, συστάσεις μας ήταν να προχωρήσουν σε νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σύντομα θέλω να αναφερθώ και στο ζήτημα της γνώσης η γνώση έχουν οι αρμόδιες αρχές των εκλογών, ε, τι δυνατότητα έχουν να προσελκύουν εμπειρογνώμονες αλλά και παρατηρητές εκλογών που να γνωρίζουν τα πράγματα. Όλο αυτό το θέμα των δεδομένων και της τεχνολογίας χρειάζεται διαφορετικά προσόντα πέρα από το να έχει πρόσβαση στα συστήματα. Δηλαδή, ποια χώρα θα πρόσφερε πρόσβαση στα πιο ευαίσθητα δεδομένα και συστήματα σελοδαπούς. Ε, ακόμα συζητούμε τι ενδεχομένω να έχει συμβεί στι εκλογέ του 2016 στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αν αναρωτηθούμε έτσι φωναχτά, εγώ ω Ευρωβουλευτή ε, αποστολή ε, παρατήρηση εκλογών, αν ζητούσα από τι Ηνωμένε Πολιτείε πρόσβαση ε, στα δεδομένα εκεί που τους χάκαραν. Θα μας έλεγαν μάλιστα περάστε ε, προς όφελος της εκλογικής διαδικασίας και της ακαιρεότητας ή θα μας έλεγαν ότι είναι ευαίσθητα τα δεδομένα οπότε δεν μπορεί κάποιος τρίτος να έχει πρόσβαση τουλάχιστον πλήρη, μάλλον περιορισμένη. Λοιπόν, τίθεται το θέμα αυτό, ποιος έχει πρόσβαση, ποιος θα πρέπει και σε ποιο πλαίσιο ε, και πάλι στην παρατήρηση των εκλογών. Αυτά μπορούν να τα γράφουν τα μνημόνια και διάφορες ε, συμφωνίες. Πολύ νωρίς όμως τη διαδικασία, όταν ακόμα δεν έχει φτάσει η αποστολή παρατήρησης, ή τουλάχιστον στο σύνολό της. Υπάρχουν κάποια άλλα σχετικά θέματα που θέλω να αναφέρω. Όσο αυξάνεται χρήση της κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε πόσο εύκολα μπορεί να κυκλοφορήσει και σε ευρύτατη κλίμακα μια ρητορική μίσους. Ε, και επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διαφήμιση με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλέξει από τους χρήστες και στοχεύουν πάρα πολύ. Ας πούμε, Μπορεί να είναι διαφορετική η ε, διαφήμιση που παίρνω εγώ, τα στοιχεία που ε, υπάρχουν στη δική μου σελίδα και σε σχέση με κάποιο άλλο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τα δεδομένα που κάποιο έχει ε, χρησιμοποιήσει. Και γίνεται πολύ στοχευμένη η διαφήμιση, και όχι μόνο στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Και στο Messenger, ας πούμε, στο WhatsApp και άλλες εφαρμογές υπάρχουν κλειστές ομάδες χρηστών, όπου είναι ακόμα λιγότερη διαφάνεια όπου κυκλοφορούν διάφοροι ισχυρισμοί και φήμες και πάρα πολύ γρήγορα διαδίδονται όλα αυτά. Και είναι δύσκολο να διαλυθούν και να, να διαψευστούν. Μερικά σχόλια τέλος για την πάρα πολύ σημαντική έννοια της εμπιστοσύνης. Στη Κένια ήλπιζαν αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη να αντικατασταθεί από την τεχνολογία. Ε, αυτό δεν γίνεται και το διαπιστώσαμε ειδής όμαση. η τεχνολογία δεν θα πρέπει να θεωρείται απομονωμένη. Υπάρχουν τα ευρύτερα ζητήματα της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, εμπιστοσύνης στους νόμους και μια σειρά από άλλα θέματα που παίζουν ρόλο. Το είδαμε και πάλι αυτό στην Κένια. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η δυσπιστία, η καχυποψία, μεγάλη υπόλωση ε, ανάμεσα στους πολιτικούς φορείς αλλά και στους θεσμούς και εντός των θεσμών, όχι μόνο μεταξύ των θεσμών. Δολοφονήθηκε και ο ειδικό πληροφορικής, ο Κρίσμα Σάντο, της ε, Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και αυτό βάρινε πάρα πολύ, ε, επισκίασε τις ε, εκλογές. Και ήταν πραγματικά στην όλη εκλογική διαδικασία ένα από τα πιο μελανά σημεία. Ακούσαμε και ισχυρισμού για hackers, για, για δεν έχουμε στοιχεία έτσι που να το τεκμηριώνουν αυτό. Αλλά και να είχαμε και να δεν είχαμε παληθεύσει πάλι δεν θα μας πίστευαν. Ε, Ήταν ε, κατάφορη αυτή η πόλωση που διέτρεχε όλη την κοινωνία και τα θέματα πληροφορικής. Σταματώ εδώ. Προσπάθησα να σας δώσω έτσι, επιγραμματικά τις ανάγκες και τα προβλήματα και πώς ε, οι νέες τεχνολογίες ε, εμποδίζουν ή δυσκολεύουν την εκλογική διαδικασία, αλλά δεν θα πρέπει να χάνουμε και τη γενική εικόνα. Το θέμα της εμπιστοσύνης είναι θεμελιώδες. Με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να ακούσω τις αποθετήσεις των άλλων μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Μαρίτε. Και τώρα να στραφώ στην Τάνια. Ένα από τα σημεία που ανέφερε η Μαρίτια ήταν ότι πρέπει να δούμε τώρα με μεγάλη προσοχή τη διαχείριση των ε, δεδομένων, την πρόσβαση, την προστασία τους και πώς αυτά μπορούν να σχετίζονται με εκλογικές διαδικασίες. Ξέρω ότι ο, ο ΑΣΕ και ο ΔΙΡ έχουν κάνει ήδη πολλή δουλειά για να αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες και να οδηγήσουν, να, έχουν, να πρωτοστατήσουν στην δουλειά αυτή για την ε, ψηφιακή διάσταση της παρατήρησης των εκλογών. Πώς θεωρείς ότι αυτό μπορεί να γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Πόσο πρέπει να αλλάξουμε τη μεθοδολογία μας από τα παραδοσιακά μέσα για να καλύψουμε και την ψηφιακή διάσταση. Ιδίω ό,τι αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα και την προστασία της ακεραιότητας των ε, ατόμων. Τάνια, ευχαριστώ πολύ. Μου άρεσαν πολύ αυτά που είπε Μαρίτια, με την ε, άμεση εμπειρία που είχε και τα απορίσματα της ήταν ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι συγκλίνουν με όσα έχω ζήσει κι εγώ. και την τροπή που έχει πάρει η μεθοδολογία του ΟΝΤΙΡ. Θα συνεχίσει και θα συνεχίσει να προσπαθεί να προσαρμόζεται όπως κάνει ήδη. Για το θέμα της πληροφορικής επικοινωνίας και τεχνολογίας, τα γνωστό ICT και τα νέα μέσα. Το βλέπετε και στο υλικό που σας μοιράστηκε, ότι σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες έχουμε πλέον κάποια έστω περιορισμένη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων. Ιδίω στην ε, ρήψη της ψήφου και την ε, ε, καταμέτρηση. Αυτά συνάδουν και με τις δεσμεύσεις σπουργονόασια και άλλες χάρτες δημοκρατικών δικαιωμάτων πρώτες εκλογές παρατήρηση εκ μέρους του Ντίρταν και του ΑΣΕ ήταν στην Εστονία. Η Εστονία, όπως θα ξέρετε, είναι η πρωτεύουσα, η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει εφαρμόσει πλήρως τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες στο εκλογικό της σύστημα. Και αρέσει σε όλους αυτό. Ωστόσο, είχαμε και δύο εμπειρογνώμονες πληροφορικάριους ε, για το θέμα αυτό που μας υποστήριξαν και συνέταξαν το μεγαλύτερο μέρος της εκθεσής μας. Νομίζω ότι ως τώρα ο Ντύρ έχει παρατηρήσει σε 14 χώρες τη χρήση των νέων ε, εκλογικών ψηφιακών μέσων σημαντικό και έχουμε πλέον έναν σεβαστό όγκο συστάσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση των ε, τεχνολογιών για τις εκλογές ε, δημιουργεί δυσκολίες στους παρατηρητές. Τα τεχνολογικά αυτά μέσα πολλές φορές χρησιμοποιούνται ώστε η άμεση παρατήρηση να γίνεται λίγο δυσχερή με σχεδόν αδύνατη. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Ωστόσο, Βάσει της εμπειρίες μας από το 2013 εκδώσαμε ένα εγχειρίδιο για την παρατήρηση των νέων ψηφιακών εκλογικών μεθόδων. Όταν τα αντιμετωπίζω και εγώ η ίδια συνειδητοποιώ ότι πρέπει να κάνω τις ίδιες δουλειές με αυτές που ισχύουν και στα επιχάρτου, στις επιχάρτου και τις, ε, τις εκλογές με υλικά μέσα. Οπότε τα ίδια πρότυπα πρέπει να ισχύουν. Πρώτα απ' όλα μυστικότητα με ένα σύστημα που ίσως θα επιτρέπει να γίνεται ηλεκτρονικό login και να ε, βλέπει ο ψηφοφόρος εάν θα υπάρχει απόλυτη μυστικότητα ή όχι. Μετά, ε, ε η κυριότητα των αποτελεσμάτων δεν δηλαδή θα πρέπει να μπορεί κανείς να εξασφαλίσει την ε, εγκυρότητα των ε, ψήφων. Ε, μετά η καθολικότητα και η οικουμενικότητα θα πρέπει να είναι το δικαίωμα αυτό προσβάσιμο σε όλους. Θα πρέπει να μπορούν όλοι να ε, έχουν τις τεχνολογικές δυνατότητες. Διαφάνεια, να υπάρχει δυνατότητα παρατήρηση, αλλά η παρατήρηση να έχει και κάποιο νόημα, λόγω χάρη το να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά ψηφοφόρων ή εξωματούχων ή υπαλλήλων με μηχανήματα που δεν λειτουργούν δεν έχει νόημα. Θα πρέπει όλοι να έχουν οδηγίε για τη χρήση των ε, συστημάτων μαζί με τα συστήματα πιστοποίηση και τα αποτελέσματα των δοκιμών. Η λογοδοσία με, με επαληθεύσιμου ελέγχου. Όπω είπαν όλοι, είναι σημαντικός, σημαντική εμπιστοσύνη του κοινού. Εάν υπάρχει επίπεδο, ένα σημαντικό επίπεδο καχυποψία, έλλειψη εμπιστοσύνη στο κοινό, τότε ε, χάνεται και η αξιοπιστία των εκλογών. Αυτό ήταν κάτι που παρατήρησαν πολλοί ε, παρατηρητές. Χρειάζεται γενική συνένεση γιατί έχει πραγματική χρησιμότητα μαζί με την δοκιμασία και την επιδίωξη της πλήρους διαφάνειας για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού. Εάν η τεχνολογία είναι μαύρο κουτί όπως αναφέρατε, λέτε ένα μαύρο κουτί δεν μπορεί να παρατηρηθεί, να είναι αντικείμενο παρατήρηση σε, μια, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με τους εμπειρογνώμονες για τις νέες εκλογικές ε, μεθόδους, τις ψηφιακές, έχουμε πλέον κάποια πείρα από τις αποστολές μας, του ΟΑΣΕ και του ΟΝΤΙΡ, και ένας εμπειρογνώμων συμμετέχει αυτή τη στιγμή στην ε, περιορισμένη αποστολή, της οποίας είμαι επικεφαλής της ε, ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο των Ηνωμένων θα είναι πολύ χρήσιμη η συμμετοχή του εκεί. Τώρα για το θέμα των κοινωνικών μέσων θα πρέπει να πω ότι ο ΟΝΤΙΡ δεν έχει ακόμα μεθοδολογία εγχειρίδιο. Κάτι το οποίο το επεξεργαζόμαστε. Χρήση του ίντερνετ στις ε, προεκλογικές εκστατείες. Υπάρχει σημαντική εμπειρία στην πράξη, την οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε σε κάποια άλλη φάση, ίσως εάν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Να στραφώ τώρα στον Ήβλιο Τέγμα. Ο οργανισμός του οποίου είστε, ο IDEA, παίζει μεγάλο ρόλο στην ε, ανταλλαγή ε, γνώσης για τις δημοκρατικές διαδικασίες, ε, τις συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες, την εκπροσώπηση. Ακούσαμε ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο κατά και γύρω από τις εκλογές. Εσείς ως πολιτικός και τώρα ως επικεφαλής του IDEA πώς ε, αποτιμάτε τις ε, δυνατότητες αλλά και τις δυσχέρειες που προκαλεί η πληροφορική. Ποιες μπορεί να είναι οι βασικές αρχές με βάση την εμπειρία σας που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν ε, εντάσσουμε την ψηφιακή διάσταση στις εκλογικές διαδικασίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και θέλω φυσικά να χαιρετήσω το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΔΕΦΚΟ, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο πρωτοπόρος παγκοσμίω όσον αφορά την ποιότητα και ακεραιότητα των εκλογικών διαδικασιών. Κοιτάξτε, πολλά μπορώ να πω για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Για να την περιορίσω κάπως. Να απαντήσω σε συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, διαχείριση τη εκλογική διαδικασία, αυτή καθ' αυτή. Δεύτερον, προεκλογική εκστρατεία και επικοινωνία. Και τρίτον, αν και συμφωνώ με του προηγούμενου ομιλητέ, κάτι που δεν έχει φύγει ακόμη, όπου μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο η πληροφορική, είναι η χρηματοδότηση των πολιτικών εκστρατιών, κομμάτων, υποψηφίων. Τι δυνατότητες έχει η πληροφορική αν αξιοποιηθεί σωστά σε όλα αυτά. Πρώτον, πληροφορική στη διαχείριση της εκλογικής διαδικασίας. Υπάρχει αυτή η αποκοπή που βλέπουμε και σε άλλους τομείς, ε, κοινωνικές σχέσεις, οικονομία. Αυτή η χρήση νέων τεχνολογιών σημαίνει ότι έχουμε τεράστιες εξοικονομήσεις και για την ε, γραφή στους εκλογικούς καταλόγους και ε, για την ίδια την εξαγωγή της ψηφοφορία και για την καταμέτρηση. Και είμαστε ακόμη σε αρχική φάση. Ίσως δεν θα χρειάζεται οι δημόσιες αρχές να επενδύουν σε μηχανήματα, αλλά μόνο σε λογισμικό. Οι ίδιοι ψηφοφόροι ή άλλες αρχές θα επενδύουν σε μηχανήματα. Είναι πολύ πιο φτηνό να ψηφίζεις ε, στο ίντερνετ παρά να ψηφίζεις ε, με χαρτί και ίσως είναι και καλύτερη προσβασιμότητα. Η ίδια η καταχώρηση στους εκλογικούς καταλόγους, ε, η ψηφοφορία και η καταμέτρηση. Όλα αυτά μπορεί να είναι και πιο διαφανή, ταχύτερα, πολύ ευχερέστερα. Αυτά είναι πολύ θετικά. Όπου αν έχουμε και περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών και βελτίστων πρακτικών μπορούμε να επιτύχουμε ακόμη πολύ περισσότερα. Και μπορούμε να αποφύγουμε και καλύτερα την νοθεία, γιατί υπάρχει λιγότερη παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Άρα μπορεί να έχουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Πολύ θετικό και αυτό για αυτές τις νέες δημοκρατίες, όπου συχνά δεν εμπιστεύονται τις δημόσιες αρχές και θεωρούν ότι υπάρχουν ε, προσπάθειες επηρεασμού των χειροκινήτων διαδικασιών. Αλλά, επίσης σημαντικό, μπορούμε να αυξήσουμε και τη συμμετοχή στις εκλογές, γιατί θα είναι πιο εύκολο να ψηφίσει κανείς. Δεν χρειάζεται να πας σε εκλογικό τμήμα, για παράδειγμα. Μπορούμε να έχουμε πολύ πιο αποκεντρωμένα κέντρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Δεν χρειάζεται να πας σε ένα κεντρικό. Και αυτό μπορεί να αυξήσει την συμμετοχή. Αλλά όπως όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες υπάρχουν και πολύ σημαντικά μειονεκτήματα. Υπάρχει πραγματική ή ε, θεωρητική ε, δυνατότητα νοθείας. Αν δούμε την αντίληψη που έχουν τα άτομα. Η θεωρητικη δυνατοτητα νοθειας αν δουμε την αντιληψη που εχουν τα ατομα η χρηση της προφορικής της εκλογικές διαδικασίες ίσως πρέπει να αντιμετωπίσει περισσότερες αμφισβητήσεις από ότι η παλιά διαδικασία. Αυτό μπορεί να είναι αντιφατικό με αυτό που είπα προηγουμένω. Κοιτάξτε. Η εμπιστοσύνη ε, κερδίζεται πιο δύσκολα από τη συμμετοχή. Και αν χάσεις την εμπιστοσύνη, ξέρεις ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να την ανακτήσεις. Η γενικευμένη χρήση της πληροφορικής, για παράδειγμα, μπορεί να εξαιρέσει την, ε, να εμποδίσει καλύτερα την ε, συμμετοχή ορισμένων. Ορισμένοι έχουν ε, πεπαλαιωμένες αντιλήψεις. Η μητέρα μου, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να εξοικειωθεί με τη χρήση πληροφορική. Την ε, επόμενη Κυριακή έχουμε αυτοδιοικητικέ εκλογές στην χώρα μου και την Παρασκευή θα πάω να πείσω τη μητέρα μου ότι μπορεί να ψηφίσει. Καλά μπορεί να μα δεσκεδάζει αυτό ορισμένου, αλλά βεβαίω και αυτοί πρέπει να ψηφίζουν και ίσως υποτιμούμε τι τμήμα του πληθυσμού έχει προβλήματα με τη χρήση πληροφορική για τέτοιου τύπου διαδικασίες. Επίσης υπάρχει ενδεχόμενο hacking και άλλα θέματα κυβερνοασφάλειας. Οπότε, θεωρώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια όχι ολοκληρωτική χρήση πληροφορικής. Να υπάρχει, για παράδειγμα, και ε, δίπλα μια καταγραφή σε χαρτί του τι γίνεται, όπου να μπορούν να δουν τα άτομα ότι βεβαίως κατεγράφει η ψήφος μου. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τη δυσπιστία που πολλοί έχουν. Τώρα, για την προεκλογική εκστρατεία, για την ενημέρωση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν. Ας δούμε πρώτα τα θετικά. Και εδώ οι νέες τεχνολογίες όχι απλά έφεραν τα πάνω κάτω για το πώς δημιουργούμε και ενημερωνόμεθα, πώς δημιουργούμε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες, είναι πολύ πιο προσβάσιμες πληροφορίες, πολύ πιο εύκολα μπορώ να ενημερώσω και να ανταλλάξω πληροφορίες με τους πάντες ε, παντού στον κόσμο. Μπορούμε να απευθυνθούμε απευθείας ε, στους υποψηφίους, στους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων. Μπορούμε να έχουμε περισσότερη επικοινωνία. Και αν εφαρμόσουμε αρχές ε, ανοιχτών τεχνολογιών, μπορούμε να έχουμε πιο διαφανείς προεκλογικές εκστρατείες και να είναι πιο προσβάσιμη η πληροφορία σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Υπάρχει λοιπόν ε, κάτι το πολύ σημαντικό και πολύ θετικό μέσω της χρήσης των ε, κοινωνικών μέσων δημιουργεί συνθήκες ε, ισότιμου ανταγωνισμού για όλους τους υποψηφίου φθηνότερο, είναι πολύ πιο φθηνό για κάθε υποψήφιο να επικοινωνήσει. Δεν πρέπει να το υποτιμούμε αυτό. Και είναι πιο εύκολη και η επικοινωνία μεταξύ πολιτών, εκλογικών αρχών και μέσων. Αλλά υπάρχουν και μειονεκτήματα. Υπόθηκαν αυτή οι λεγόμενοι ε, χώροι ε, αντίχησης, η κατάχρηση, οι επιθέσεις μέσω bot. Το μόνο που θέλω να προσθέσω, με βάση την πείρα που έχουμε, θεωρούμε ότι η αυτορύθμιση που, ζητάει, που ζητούν οι μεγάλοι ε, επιχειρηματικοί όμιλοι Google, Apple, Facebook και Amazon δεν αρκεί. Πρέπει οι δημόσιες αρχές και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξουν το σημαντικό τους ρόλο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μειονέκτημα. Σε σχέση με τη διαφάνεια. Παρά το ότι έχει αυξηθεί πολύ διαφάνεια, μειώνονται τα θέματα του ιδιωτικού βίου οι υποψήφοι ασχολούνται με την κατάσταση μόνο των ψηφοφόρων, αλλά ένας υποψήφιος σε τι πιέσεις μπορεί να εκτεθεί. Πόσα στοιχεία από την προσωπική σου ζωή πρέπει να τα κοινοποιήσει. Στην Ινδονησία ένας νέος κανονισμός λέει ότι οι υποψήφοι πρέπει να γνωστοποιούν τις ιατρικές τους πληροφορίες. Είναι σημαντικό και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό η πληροφορική δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προεκλογική στρατεία και τις ροές ε, ενημέρωσης μεταξύ δημοσίων αρχών, εκλογικών αρχών, ψηφοφόρων και υποψηφίων, αλλά και τη χρηματοδότηση όλου του εκλογικού οικοσυστήματος. Έχει αλλάξει ριζικά. Υπάρχουν ορισμένα θετικά. Για παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση από του ε, ψηφοφόρου. Πριν από 12 χρόνια ο Μπαράκ Ομπάμα, Ομπάμα ξεκίνησε να συλλέγει χρήματα μέσω του διαδικτύου. Έτσι εξισώνονται οι συνθήκε ανταγωνισμού των υποψηφίων σε σημαντικό βαθμό. Η σωστή χρήση πληροφορικής και ίντερνετ μπορεί να κάνει πιο ευρέως γνωστές και κοινοποιήσιμες τις πηγές χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατιών. Αυτό σημαίνει περισσότερη διαφάνεια. Άρα να μειωθεί ο κίνδυνος διαφθορά. Έχουμε εργαστεί πολύ σε αυτά. Έχουμε κάποια εγχειρίδια, δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Ωστόσο πρέπει επίση να πούμε ότι και εδώ πρέπει κάπως να διαφοροποιήσουμε τα πράγματα. Κάποια συστήματα που καθιστούν πιο εύκολο να αποκαλυφθούν οι πηγές χρηματοδότησης κάποιων εκστρατιών, τα συστήματα αυτά είναι ακόμη εθελούσια ή πειραματικά μόνο ε, αν τα συστήματα είναι επαρκώς ψηφιακά όρημα μπορούν να είναι αποτελεσματικά, αλλιώ μπορεί να γίνουν καταχρήσεις. Οπότε υπάρχουν τα υπέρ αλλά και τα κατά. Και για τη διαχείριση των εκλογικών διαδικασιών και τον τρόπο διεξαγωγής των προεκλογικών εκστρατιών και τον τρόπο που επι, επικοινωνίας μεταξύ εκλογικών αρχών και πολιτών υπάρχουν υπέρ και κατά και τρίτον αυτή η γνωστοποίηση πηγών χρηματοδότησης και ο έλεγχος των ε, οικονομικών ροών προς τους υποψηφίους και τα κόμματα και εδώ πολλά πρέπει να κάνουμε παραπάνω και μπορούν να γίνουν με την ε, επέκταση της χρήσης της πληροφορικής. Ευχαριστούμε πολύ. Μια πρακτική παρατήρηση. Μου είπανε ότι όσοι θέλετε να μιλήσετε μετά για να κάνετε κάποιο σχόλιο μια ερώτηση, έχετε μπροστά σας ένα μικρό φύλλο χαρτί που μπορείτε να το συμπληρώσετε, ένα δελτίο. Δεν είναι εγγραφή με την έννοια που χρησιμοποιούμε στην πληροφορική. Απλώ μπορούμε να δούμε πού κάθεστε, ε, κυρίω για τον αριθμό του εδράνου και για να μπορώ να σα δώσω εγώ το λόγο στη συνέχεια. Σα προσκαλώ λοιπόν να συμπληρώσετε το έντυπο, αν έχετε σχόλια και ερωτήσει. Και τώρα, με την ε, μακρά σου εμπειρία στην ε, παρατήρηση εκλογών. Έχεις δει να γίνεται όλο και πιο ψηφιακό το περιβάλλον και στη διάρκεια του, ε, των εκλογών και με την παρατήρηση και στην προεκλογική εκστατεία. Ποια είναι η άποψή σου λοιπόν για την όλη μεθοδολογία και στην ευρωπαϊκή μεθοδολογία ένα σημαντικό στοιχείο είναι να παρακολουθούμε εκλογές και το πώς προβλήθηκαν στα μέσα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ότι τι γίνεται και στα κοινωνικά μέσα, στα κοινωνικά δίκτυα. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Όπως είπε και η Μαρίτια, ποιες είναι οι ελάχιστες εγγύσεις που μπορούμε να ζητήσουμε από τη χώρα υποδοχής ως προς την πρόσβαση τις αποστολής παρατήρησης των εκλογών και τον τρόπο που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να επηρεάσουν την ε, αγκαιρεότητα και την διαδικασία. Το πρώτο που θα κάνω είναι να σας ε, δείξω έναν τεράστιο καθρέφτη για να μπορέσετε όλοι να δείτε τους εαυτούς σας μέσα διότι ξέρω ότι ο καθένα και κάθε μία από εσά έχετε συμμετάσχει σε πάνελ και έχετε υπάρξει τελευταίο ομιλητή. Και ξέρετε ότι όταν φτάσει η σειρά σα, όλα που πρέπει να πει κανεί έχουν ήδη καλυφθεί από του προηγούμενου. Τι συμβαίνει λοιπόν, έχει κανεί τεράστια ελευθερία ω τελευταίο ομιλητή. Μπορεί να παραμείνει σιωπηλό και να πει πάμε απευθεία ερωτήσει, αλλά παρά είναι πολλοί αυτοί στο ακροατήριο που με γνωρίζουν. Εγώ δεν ε, αφήνω ανεκμετάλλευτε τις ευκαιρίες να παραμείνω σιωπηλό. Γι' αυτό θα πάω ένα βήμα πιο πίσω και θα ε, ακολουθήσω την πρόταση του Πρόεδρου Ταγιάννη να ε, είναι η συζήτησή μας αυτή αμφίδρομη και να σεβαστούμε τη δημοκρατία και του κυρίου παντζέρι που είπε να θέσουμε το όλο ε, θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Διότι το να μιλάμε για τεχνολογικά μέσα χωρίς να καταλαβαίνουμε το ε, είναι οι υπηρεσίες, ποιες είναι οι υπηρεσίες για τις οποίες εκτελούμε τα διάφορα, τις διάφορες διάφορα καθήκοντά μα, ποιες είναι οι αρχές, οι νομικέ αρχές βέβαια των οποίων δρούμε, τότε χάνουμε λίγο και την ουσία της δουλειά μας. Θέλω λοιπόν και για όσους με γνωρίζετε δεν θα βάλω τώρα το καπέλο του καθηγητή νομικής για να μιλήσω για αυτά τα θέματα με αυτόν τον τρόπο αλλά αυτό το γεγονός με το οποίο έρχομαστε αντιμετώπιση συνεχώς είναι το εξής αν μιλάμε για λαϊκή βούληση και λαϊκή κυριαρχία, μιλάμε για λαό, για έθνος. Η κυβέρνηση που μπορεί να επισκεπτόμαστε και μας έχει προσκαλέσει, μπορεί να έχουμε πάει και από μόνοι μας, ε, ε, διενεργεί μια πράξη ουσίας που είναι θεμελιακή αν θέλει να είναι η χώρα δημοκρατική. Ε, εκλογές ε, αδιάβλητες εκ μέρους των πολιτών είναι ουσιαστική πράξη για να εξασφαλίσει την νομιμοποίησή της και για τους ενώπιον των πολιτών της, αλλά και για το πώς εντάσσεται στο ευρύτερο διεθνές ε, προσκήνιο, την ομάδα των εθνών, των κρατών του κόσμου. Για να το πω με απλό τρόπο, οι εκλογές είναι του λαού, του κόσμου. Ό,τι κάνουμε στον κόσμο μας, τα πρότυπα που θέλουμε να προωθήσουμε, οι μεθοδολογίες που θέλουμε να καλλιεργήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε, όλα αυτά πρέπει να απορρέουν από αυτή τη βασική κατανόηση. Και ω διεθνεί φορεί πρέπει να παρακολουθήσουμε, να συνοδεύσουμε την όλη διαδικασία αυτή. Δηλαδή πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο πολίτη μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασίες που δίνει την εμπιστοσύνη ότι οι εκλογές είναι γλύσει και διάβλητες. Όχι μόνο εκλογές που πρέπει να είναι διάβλητες και ανώθευτες, αλλά ε, να γνωρίζει ο κόσμος, ο ψηφοφόρος, ότι οι εκλογές αυτές ε, δεν ε, νοθεύτηκαν. Ε, διότι η λαϊκή εμπιστοσύνη είναι τυφλή. Αν ο κόσμος δεν βλέπει τις διαδικασίες και δεν μπορεί να τις πιστέψει, θα έχει καχυποψία. Αυτό υπονομεύει την διεξαγωγή των εκλογών και την ανάληψη της εξουσίας που είναι νόμιμη και φιλελληνική. μπορεί να δώσει έναυσμα για πράξεις βίας, για αμφισβητήσεις. Αυτό κινητοποιεί τον κόσμο για να αντιδράσει. Ε, πήγα μετά τη Μαρίτια στην Κένια και πήγα με την Μαρίτια στην Κένια και είδαμε όχι πρόβλημα με τα ψηφιακά, αλλά κατανοησία. Δεν μπορούσε ο κόσμος να καταλάβει πώς πρέπει να λειτουργήσει σωστά η διαδικασία και να την φέρει εις πέρα σωστά. Διότι το πρόβλημα δεν είναι τα αποτελέσματα των εκλογών τα ανακριβή. Ήταν κανεί δεν πίστευε τα χάρτινα ψηφοδέλτια και την καταμέτρησή του. Υπήρχε ανικανότητα να ε, αποδείξει κανείς την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Μέρος του προβλήματος ήταν ότι υπήρχαν συμβάσεις ιδιοκτησίας με ξένες εταιρείε όπου ε, τα, ο βασικός όγκος των πληροφοριών και των δεδομένων είχαν πάει εκτός της χώρας. Άρα δεν μπορούσαν νομίμως να αποκαλυφθούν ώστε εγκαίρω το δικαστήριο να έχει επίγνωση της φύσης της διαδικασία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια από τι θεμελιώδει αντιφάσει από τα, αμφιλεγόμενα, από τα ε, παράδοξα που έχουμε αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να δούμε κατά πόσο οι διαδικασίες της Κένια ή άλλων χωρών είναι, επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων, ε, αν είναι διαφανείς και αν επιτρέπουν τη δημιουργία της λογοδοσίας. Εδώ μας ενδιαφέρει να δούμε αν υπήρχε κοινοβουλευτική παρακολούθηση, νομική παρακολούθηση, αν είχαν τη δυνατότητα τα κόμματα και οι πολίτες να έχουν γνώση των αποφάσεων βάσει των οποίων οι τεχνολογίες θα έλυναν το πρόβλημα που αποτελούσε πρόβλημα στην Κένια. Ήταν κάτι που προσπαθούσαν κάποιοι με κάποιους ειδικού πληροφορικής ή ε, κάποια στελέχη της κυβέρνησης προσπαθούσαν να κάνουν μια αγορά εκ μέρους κάποιων. Εκεί είναι μια διάσταση που ίσως παραγνωρίστηκε. Το θέμα δεν επικεντρώθηκε λοιπόν στην ημέρα των εκλογών, αλλά στα προηγούμενα στάδια. Δηλαδή ακόμη και πριν την ε, μακροχρόνια παρατήρηση των εκλογών, όπως την έχουμε ονομάσει. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να κοιτάμε την πολιτική διαδικασία και όχι μόνο τη διενέργεια των εκλογών. Αλήθεια είναι και αυτό. Αλλά όσοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τέτοιε διαδικασίε βρίσκονται στη χώρα ούτω ή άλλω. Οπότε, ε, όπω ξέρετε, όλοι οι πολιτικοί θύνοντε στην αίθουσα αυτή όσοι είστε, η ευρωπαϊκή πολιτική, πιστεύω ειστε η ευρωπαικη όπω και η διατλαντική πολιτική, θα πρέπει να στραφεί στο να ενθαρρύνει τι αρχέ τη συμμετοχή όλων, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Θα πρέπει αυτά να εφαρμόζονται και όταν καλούνται κάποιοι να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά μέσα, το ίδιο και για τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά θα το θίξω για αυτό το θέμα κάποια στιγμή ξεχωριστά. Νομίζω λοιπόν ότι το να ξεπεράσουμε το μαύρο κουτί που ανέφερε και η Ματιά είναι κρίσιμη σημασία. Θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Αμερικανική ε, Υπηρεσία για την Διεθνή Ανάπτυξη, γιατί θέλετε να χρηματοδοτήσετε την αγορά τεχνολογικών μέσων και εργαλείων που δεν έχουν λάβει υπόψη τους αυτές τις αρχές ε, ούτως ή άλλως, εξ αρχής. Μιλάμε για διεθνή πρότυπα. Διεθνή πρότυπα που προκύπτουν από τον ΟΗΕ και τα εργαλεία του, από όλες τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από από όλου όσοι ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε περιοχή του κόσμου, από σχετικέ διακηρύξει και ανακοινώσει που ανέφερε και οι, υπογραμματέα, οι γενικοί υπογραμματές και θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί να αγοράσουμε αυτά τα τεχνολογικά μέσα εάν δεν υπάρχει απόφαση συμμόρφωσης και εάν αυτή η τεχνολογία δεν καλύπτει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και από αυτή τη σκοπιά την παρατήρηση των εκλογών. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι πολίτες πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν ότι οι εκλογέ τους είναι αδιάβλητε, ε, Θα πρέπει να έχουν κρίσιμε πληροφορίε στα χέρια τους. Ε, η Μαρίτια το είπε και αυτό. Εάν δημιουργήσουμε νέους ε, καταλόγους, ας πούμε, ψηφοφόρων, βιομετρικούς, τι θα γίνει με την αποστολή των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα αυτά είναι πολύ εύκολο να τα έχει κάνει αμέσω. Και η αρχή των ανανεχτών δεδομένων που ανέφερε και ο Ιβ είναι ε, εύκολο να εφαρμοστεί στην εκλογική διαδικασία. Τα ανοιχτά δεδομένα θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα αμέσω και με τρόπο που να είναι και έγκαιρο δηλαδή μπορεί κανείς να επαληθεύσει αμέσως τα αποτελέσματα. Στη Ζιμπάμπουε έγινε αυτό, ήδη, μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη φορά. Το αποτέλεσμα όμως θα πρέπει να διατίθεται η τελεσπόδο κατάλογος των ψηφοφόρων εγκαίρω, αμέσως και με τρόπο ε, τεχνικής λεπτομέρεια, δηλαδή να είναι γνωστά τα πάντα. Θα πρέπει να είναι πλήρη, να είναι ε, δωρεάν και διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Υπάρχουν και άλλε αρχέ που έχουμε αναπτύξει στην δική μας ε, την ε, οργάνωση, στο NDI. Δεν υπάρχει χώρα που να μην μπορεί να το σε αυτά τα πρότυπα. Άρα η απάντηση στην ερώτησή σα είναι ναι, υπάρχουν βασικά πρότυπα και τα επεξεργαζόμαστε εδώ και αρκετό καιρό. Και ένα ακόμη σημείο για το κομμάτι της πληροφορικής, το οποίο και πάλι κάποιος το επενήχθηκε. Διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης του, της διαδικασίας του δημόσιου διαγωνισμού. Εάν δεν μπορεί κανείς να δει πώς ελήφθη η απόφαση και τι έγινε εφόσον η η απόφαση, δηλαδή ότι το τεχνολογικό μέσο σκοπό έχει αναλύσει ένα πραγματικό πρόβλημα που έχει εντοπιστεί από κάποιου, ποιε είναι οι τεχνικέ προδιαγραφέ, καλύπτονται, έχουν γίνει τα τεστ κοπόσεω και όλα τα σχετικά που απαιτούνται. Αυτά είναι μέρη μια ανεξελίξη διαδικασία θα πρέπει να είναι ανοιχτή και ε, χωρί συγκεκριμένο τέλο. Θα πρέπει λοιπόν οι εμπειρογνώμονε να μελετήσουν και τι διαδικασίε των προμηθειών. Κάτι το οποίο έχουμε να, το, σκοπό να το δούμε με κάποιε νέε τεχνικέ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Θα στραφώ εντό ολίγου και στα κοινωνικά δίκτυα. Διότι ξέρουμε ότι είναι κάτι που απασχολεί την επικαιρότητα. Και πάλι για τα κοινωνικά δίκτυα, όταν μιλάμε για εκλογέ και μιλάμε για τον εκλογικό κύκλο. Οι εκλογέ δεν είναι μόνο η μέρα τη ψήφου, αλλά είναι μια σειρά από διαδικασίε που προηγούνται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το επόμενο βήμα το επόμενο βήμα είναι ότι οι εκλογέ μπορούν να διαχωριστούν. Δεν μπορούν να διαχωριστούν το πολιτικό και το κοινωνικό ιστό μια χώρα. Το θέμα των κοινωνικών μέσων και τη πληροφορία, τη αγκαιρότητα τη πληροφορία και τη παραπληροφόρηση, το αποδεικνύουν με τρόπο ανάγλυφο. Οι πολίτε θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ε, κάνουν την επιλογή του όταν ασχολούνται με την πολιτική, όταν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν στην κάλπη δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε καταπίεση. Η επιλογή του θα πρέπει να είναι εντελώ ανεξάρτητη και ελεύθερη, αλλά θα πρέπει να είναι και τεκμηριωμένη. Τώρα, αν θέλουν να μάθουν ε, για το χαρακτήρα των πολιτικών ή για τα εθνικά ζητήματα που διακυβεύονται στι εκλογέ, ή ε, το κατά πόσον η ίδια διαδικασία των εκλογών είναι αδιάβλητη, ε, πρέπει οι πληροφορίε να είναι διαθέσιμε αμέσω. Ε, τα ανοιχτά δεδομένα είναι σημαντικά εδώ. Αυτό είναι το είδο των πληροφοριών που χρειάζονται. Α πούμε, πώ χρηματοδοτήθηκε η προεκλογική εκστρατεία του καθενό, και αυτό είναι ένα τομέα που πρέπει να ξέρουμε πώ να ερευνήσουμε. Αλλά αν οι πληροφορίε παρακρατούνται, Εάν οι πολίτες δεν μπορούν να δουν αυτές τις βασικές πληροφορίες, αυτό δεν είναι ελεύθερη, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη εκλογή. και προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο διαταραχή στην σωστή πληροφόρηση παρά παραπληροφόρηση είναι άλλο η κακή πληροφορία και άλλο διακοπή. Δηλαδή δεν ε, είναι μόνο οι ψεύτικες πληροφορίες για τον αντίπαλο κάποιου, αλλά και πληροφορίες που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα και που με την ύπαρξή τους δημιουργούν έλλειψη εμπιστοσύνης και ερωτηματικά. Αυτό από μόνο το αρκεί για να δημιουργήσει σύγχυση. Ε, υπεύθυνοι μπορεί να είναι και πολλοί και διάφοροι. Ε, οι ανταγωνιστές ή εκτός της χώρας. Τα ξέρετε καλά κι εσείς όσοι κάθεστε εδώ, ιδίω όσοι είστε από την Ευρώπη, αλλά είτε κοιτάμε τι γίνεται στην Καμπότζη, είτε σε άλλες χώρες, ας πούμε το δημοψήφισμα στην Κολομβία για την ειρηνευτική πρωτοβουλία, Εκεί υπήρχε δυσυνοριακή παρέμβαση από εξωκρατικούς ε, παράγοντες και παραπληροφόρηση. Και δεν είναι μόνο ιδεολογική για τα κίνητρα. Αυτό στην Κολομβία μπορεί να ίσχυε. Το έχουμε δει και στο Μεξικό κι αλλού. Αλλά μπορεί να είναι ε, και συνδικαλιστικές εγκληματικές οργανώσεις. Εδώ ε, πρέπει να δούμε βεβαίως το, ότι η διαφορά μεταξύ παραπληροφόρησης ε, και των άλλων μορφών είναι κάτι θα το κρίνουν οι ακαδημαϊκοί. Αλλά έχουμε και τους φίλους μας στα μέσα, μα... στα μέσα μαζικής ε, επικοινωνίας που συγκεντρώνουν τα δεδομένα τους. Έχουμε αυτούς που ασχολούνται με την κοινωνική πληροφόρηση, κοιτάζουν ε, πώς λειτουργήσε το ένα μέσο και το άλλο. Εμείς ως διεθνείς παρατηρητές Πρέπει να μάθουμε πώς να ε, αξιοποιούμε τους πόρους που παρέχουν οι παρατηρητές για τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα διεθνώς και ε, επιμέρους. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι με το θέμα αυτό ασχολούμαι εδώ και 25 χρόνια και ως παρατηρητής εκλογών διεθνώς και βοηθώντας ε, τους ε, πολίτες και τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων και όλους όσους χρειάζεται να βρουν λύσεις για τα θέματα αυτά. Στην ε, διεθνή παρατηρήση λοιπόν εκλογών θα περιοριστούμε σε ένα σημείο που θα έχουμε τόσο πολύ σκορπιστεί ε, που δεν θα μπορούμε να καλύψουμε όλες τις αποστολές που θέλουμε να κάνουμε, αλλά ε, θα έχουμε τόσο λίγες ειδικέ γνώσεις που δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε πραγματικά τις εκλογές και να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών, δηλαδή οι εκλογές τους να είναι ανεξάρτητες, αδιάβλητες και δημοκρατικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πατ. Ευχαριστώ και τους τέσσερις ομιλητές μας. Έχω πολλές ερωτήσεις εδώ, αλλά και πολλές ερωτήσεις βλέπω να έχετε κι εσείς από το κρατήριο. Θα αφήσω τις δικές μου στην άκρη λοιπόν και θα ακούσουμε τις δικές σας. Εκτός αν θέλει κάποιος από τα μέλη του πάνελ να κάνει κάποιο σύντομο σχόλιο για να περάσουμε αμέσως μετά στις ερωτήσεις ε, από το κοινό. Πολύ σύντομα η κυρία Σχάκια, γιατί έχει σημασία αυτό. Για τη συνεχιζόμενη παρατήρηση της πολιτικής διαδικασίας, το μήνυμα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς, γιατί βεβαίως θα πρέπει να δίνεται συνέχεια και να επικαλύπτεται και η παρατήρηση των εκλογών με τη μόνιμη πολιτική. Θα πρέπει συνεχώς να ε, ανατροφοδοτούνται αυτά τα δύο. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στη πολιτική διαδικασία, τη, την παρακολούθησή έτσι και την οποιαδήποτε μόνιμη πολιτική. Κοίταξα πόσο κόστησαν οι εκλογές στην Κένια. Όταν είπε ο κύριος Λετέρμο ότι θα μπορούσε να μειωθεί το κόστος, ε, στην Κένια 19 ε, εκατομμύρια ε, οι ψηφοφόροι, 500 εκατομμύρια, 25 δηλαδή ε, ε, δολάρια Ηνωμένων Πολιτείων. Ενώ στην Ιγυρία 79 εκατομμύρια πιθανή ψηφοφόροι, 630 εκατομμύρια ε, αμερικανικά δολάρια το κόστος, περίπου 8,6 δολάρια ανά εκλογέα. Το 1 τρίτο δηλαδή του κόστους. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με την πληροφορική, που δεν σημαίνει ότι η πληροφορική μειώνει το κόστος αυτόματα. Και το ε, ε, επόμενο θέμα, το μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ίση κανόνες παιχνιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πού έχω καταλήξει τώρα εγώ στη σκέψη μου. Για τα κοινωνικά μέσα βεβαίως είναι μια πλατφόρμα για να εκφράζεται το κάθε πρόσωπο. Βεβαίως υπάρχει ελευθερία της έκφρασης, αλλά ε, ε αναφέρθηκε και ο Πάτης αυτό. Ε, ότι εκείνος, εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα ε, να ε, χρησιμοποιούν με εκθετικό τρόπο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον μέσο μεμονωμένο χρήστη. Κάποιες εταιρείες Δηλαδή, όλο και περισσότερο ε, έχουμε μία αγορά, αλλά όχι με την έννοια της αγοράς όπου ανταλλάσσονται ιδέες και γίνεται πολιτική συζήτηση, αλλά της αγοράς όπου γίνεται εμπόριο. Και ποιο είναι το μήνυμα, ποιος το μεταφέρει αυτό το μήνυμα, ποιος είναι ο αγγελιοφόρος και ε, τι ε, θέλει να πει. Άρα όλα αυτά υπονομεύουν ε, το ίσους παιχνιδιού. Ευχαριστώ Μαρίτσια Και με την άδειά σας και των τεσσάρων να δώσουμε το λόγο ε, στο κοινό. Η κυρία Σέντεφερ πρώτη που κάθεται στο έδρανο παρελθόν 44. Μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου και ε, της Περιβαλλοντικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε και μοιραστήκατε τις γνώσεις σας μαζί μας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την πληροφορική. Βεβαίω, αυτή την εξέλιξη δεν θα πρέπει να τη σταματήσουμε, δεν μπορούμε και να τη σταματήσουμε, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε τι χώρε που, την ε, χρησιμοποιούν και να ε, βοηθήσουμε για άλλε. Υπάρχουν όμω πολύ κρίσιμα ζητήματα. Το ένα είναι η διαφάνεια, όχι μόνο για του παρατηρητέ και για του ψηφοφόρου, για μια κοινωνία. Πολύ συχνά όταν έχουμε παρατήρηση εκλογών και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην κοινωνία, δεν υπάρχει ευθύνη, δεν υπάρχει απόδοση ευθυνών και υπάρχει διαφθορά. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και για τα συστήματα πληροφορική και ηλεκτρονικής ψηφοφορία. Αλλιώ υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος να αυξάνεται συνεχώ η αποχή. Και όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για μια δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτό για να υποστηρίζουμε τις χώρες και να τις συμβουλεύουμε για να οικοδομούν αυτό το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με πολύ μεγάλη διαφάνεια, αλλιώς είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έλισαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο έδρανο 25. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ ε, τους διοργανωτές ε, της παρούσης διάσκεψης και τα μέλη του πάνελ γιατί πραγματικά τέτοιες διοργανώσεις βοηθούν να ανταλλάσσουμε απόψεις, βέλτιες πρακτικές και να ε, μοιραζόμαστε γνώσεις. Συγχαρητήρια λοιπόν από πλευρά μου. Και, ο κύριος Μέλο με προβλημάτισε όταν άρχισε να μιλάει για αυτό τον καθρέφτη. Έψαχνα τον αριθμό του εδράνου μου και δεν το βρήκα. Και δεν είναι αριθμό Εδράνο, είναι ε, αριθμό γραφείου. Και έπρεπε να σηκωθώ να σκύψω να δω το γραφείο μου. Οι, άλλοι ε, ίσω θα μπορούσαν να βοηθηθούν από αυτή την ε, αναφορά. Μάλιστα, πολύ χρήσιμο. Εμείς είμαστε ο καθρέφτης και σας βλέπουμε. Ε, τουλάχιστον κάτι πυροδότησα κι εγώ και έδωσα τροφή για σκέψη. Λέει ο κύριος Μέρλο. Ο κύριος Κίσεχελ πόκο από την Αφρικανική Ένωση στο έδρανο 102, δεν απατώμε. Εσείς εκεί πίσω. Παρακαλώ. Αν θέλετε μπορείτε να μιλήσετε γαλλικά, ε, έχουμε πολλές γλώσσες. Παρακαλώ. Ό,τι προτιμάτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ε, το μικρόφωνο σε αναμένω. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας εκφράσω μια ανησυχία που έχω. Για κάποιες λύσεις που θα μπορούσαμε να προτείνουμε μετά α, ε, τις ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων που είχαμε. Καλό είναι να καταγγέλουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά καλύτερο να προσπαθήσουμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις για να αποφύγουμε ε, τη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης στις εκλογικέ αναμετρήσεις της χώρας μας. Σήμερα στην Αφρική το φαινόμενο αυτό δεν ξέρουμε πια πώς να το ελέγξουμε. Ε, έχει ε, προσλάβει τεράστιες διαστάσεις και έχουμε συκοφαντίες ε, και δολοφονίες χαρακτήρων στα κοινωνικά μέσα. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή τη ροή ψευδών πληροφοριών που έρχονται να διαταράξουν καμιά φορά την εκλογική διαδικασία. Θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις εδώ και στα πλαίσια της σημερινής ανταλλαγής απόψεων. Έχουμε αυτή την απειλή λοιπόν που είναι χειρότερη από την ίδια την τρομοκρατική απειλή τη σήμερα ημέρα. Διότι έχουμε διάφορες προφορίες έτσι, με τέτοια ροή που δεν ξέρουμε ποια είναι η πηγή τους, ποια, ποιος είναι ο στόχος, ούτε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος τους ε, στις εκλογές. Αυτό είναι, αυτή είναι η ρωτά λοιπόν. Τι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. 90, Γκάιλ Μικάλεφ από την Επιτροπή Βενετία. Ευχαριστώ πολύ. Δύο σχόλια και μία ερώτηση. Πρώτο σχόλιο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε μία σύμβαση για την ε, κυβερνοεγκληματικότητα που είναι το μόνο διεθνέ κείμενο μέχρι στιγμής για το θέμα αυτό. Μπορεί να σα ενδιαφέρει. Γι' αυτό το αναφέρω. Και εργαζόμεθα και για ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο σε αυτή τη σύμβαση για, τον, για την ενημέρωσή της, ιδιαίτερα για την προστασία των δεδομένων. Δεύτερον, παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσει κατά τις προεκλογικές εκστρατείες. Ξέρουμε ότι είναι σοβαρό πρόβλημα για τις δημοκρατικές εκλογές και έχουν ως επίπτωση να μην ε, ανταγωνίζονται όλοι οι υποψήφοι με ίσες συνθήκες. Είναι μεγάλα θέματα αυτό. Ελεύθερη έκφραση, αλλά και ισότιμη συμμετοχή στι εκλογέ. Θεωρείται ότι, ότι η παραπληροφόρηση και οι ψευδεί ειδήσει τι ε, διαχωρίζω ε, ε, επί τούτου είναι τμήμα τη ελεύθερη έκφραση και πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές γιατί μέχρι στιγμής είναι σύντομοι. Σπάνιο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ντίντο Ράσο από την ε, Βουλή της Κένειας. Θέση 148. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Μαρίτια που έπαιξε ρόλο παρατηρήτρια στι εκλογέ στην Κένια. Τονίζω ευθύ εξ αρχή ότι είναι σημαντικό όλοι να καταλάβουμε ότι οι εκλογές αυτές στην Κένια ήταν έξι εκλογέ σε μία και η μόνη εκλογή η οποία αφισβητήθηκε ήταν οι προεδρικές εκλογές. Αυτές ακυρώθηκαν. Είναι σημαντικό να το ξέρετε αυτό. Θέλω να πω ότι αν πρόκειται να πάνε στις κάλπες αύριο οι πολίτες μου στην Κένια, ως ε, μέλος του Κοινοβουλίου τονίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την πληροφορική. Όχι με τον παραδοσιακό τρόπο που χρησιμοποιήσαμε στις προηγούμενες 11 εκλογές. Ενώ μόνο σε αυτή τη 12η λοιπόν χρησιμοποίησαμε την πληροφορική. Η χρήση πληροφορικής εγγυώνται περισσότερο το αδιάβλητο των εκλογών από ότι οι παλιέ ε, διαδικασίε. Γιατί πολλέ φορέ είχαν πολλά ψηφοδέλτια στι κάλπε ε, συμπληρωματικά. Το ερώτημα που θέτω λοιπόν είναι θέλουμε να διορθώσουμε την εκλογική διαδικασία ή να διορθώσουμε την πολιτική. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Επίσης, εξετάζεται εκλογές στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες. Μήπως ήρθε η ώρα και να κοιτάξουμε και τι γίνεται και στις δικές σας. Για να δούμε, δούμε εδώ τι γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει ε, ε από δίπλα ε, ένα αντίγραφο σε χαρτί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εκλογές σας ήταν αδιάβλητες. Ή Υπάρχουν ερωτηματικά. Μήπως το θέμα είναι να διορθώσουμε παντού στις χώρες μας το εκλογικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ σωστό αυτό που είπατε. Τζιν Λάμπερτ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέση 23. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, να σχολιάσω ορισμένα που υπόθηκαν. Όσοι έχουμε συμμετάσχει σε τέτοιες αποστολές, κάτι που με συναρπάζει είναι όταν επιστρέφω στη χώρα μου και διαπιστώνω ότι και εκεί γίνονται πράγματα που θα έβαζα σε έκθεση παρατήρησης λέγοντας ότι θα έπρεπε να βελτιωθούν την επόμενη φορά. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε όλοι. Αυτή η αταξία γύρω από την πληροφόρηση που αναφέρατε. Κοιτάξτε, είμαι από τη Βρετανία, καταλαβαίνετε. Ποιοι είναι οι θεσμοί που απολαμβάνουν εμπιστοσύνη όπου πιστοποιείται ότι είναι αδιάβλητοι η διαδικασία και σωστές οι πληροφορίες. Αν η Κεντρική Εφορευτική, Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να αντιδρά ταχαίω, θα βοηθούσε. Αν, για παράδειγμα, διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες, επειδή η αστυνομία απαγόρευσε τις μετακινήσεις, λέγεται ότι η αστυνομία απαγόρευσε τις μετακινήσεις. Θα έπρεπε να μπορεί κάπως, ε, κάποιος να ελέγξει. Θα έπρεπε λοιπόν οι κεντρικές εκλογικές αρχές ε, να αναπτύξουν τέτοιες δυνατότητες. Και πρέπει να επενδύσουμε και σε σωστή δημοσιογραφία. Να υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας. Οι δημοσιογράφοι να ελέγχουν τις πηγές τους πριν δημοσιεύουν ό,τι δημοσιεύουν. Σημαντικός λοιπόν και ένας κώδικας δοντολογίας. Πολλοί σχολιαστές θεωρούν ότι η τεχνική πλευρά του θέματος είναι βαρετή και δεν κάνουν αυτό που χρειάζεται ούτως ώστε να υπάρχουν και τεχνικές προφορίες γνωστές σε όλους. Και για αυτά τα κηρύγματα μίσους. Μα δεν ευθύνονται και τα κόμματα όταν υπάρχουν μέλη τους που μέσω των κοινωνικών μέσων ε, διαδίδουν τέτοια μηνύματα μίσους. Και τι κάνουν τα πολιτικά κόμματα. Για παράδειγμα, διαγράφουν κάποια μέλη, αποσύρουν την υποψηφιότητά τους ή απλώς ε, κάνουν τα στραβά μάτια και εποφελούνται από αυτές τις ψευδείς ειδήσει που κάποιοι διαδίδουν και τις οποίες κάποια στιγμή μετά θα τις διαψεύσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάριο Γκάλια από τη Μάλτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Ξέρετε ότι πολλές φορές και η παρατήρηση γίνεται ε, μέσω πολιτών της χώρας αυτής, οι οποίοι συλλέγουν και πόρους. Ορισμένοι λένε ότι αυτή η παρατήρηση μπορεί να βοηθήσει και τους διεθνείς παρατηρητές για να μάθουν τι γράφεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν υπάρχουν ε, διάφορες τάσεις ε, που φαίνεται ότι προέρχονται από, ένα συγκεκριμένο, από μια συγκεκριμένη πηγή ή αν ε, κάποιοι κάνουν ε, προπαγάνδα υπέρ βίας. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε βέβαια να υποκαταστήσουμε τις παραδοσιακές αποστολές διεθνούς, διεθνούς παρατήρησης, αλλά μέσω της συμμετοχής των πολιτών της χώρας αυτής μπορούμε να συμπληρώσουμε και να βοηθήσουμε τις ε, παραδοσιακές αποστολές παρατήρησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Φέτλινγκ από τη Διεθνή Ένωση για την Παρατήρηση Εκλογών, στην 123. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που ήταν ε, αρκετά συγκρατημένη συμμετέχοντες στο πάνελ όταν ε, μιλούσαν για τις διακοπές που μπορεί να υπάρξουν με τη χρήση των ε, μέσων της τεχνολογίας πηγαίνοντας από την, ε, τους βιομετρικούς καταλόγους ψηφοφόρων μέχρι την ηλεκτρονική ψήφο. Υπάρχει το εμπόδιο της τεχνολογίας ε, και μπορεί να υπάρχει μια προκατάληψη διότι τεχνολογικά μέσα βελτιώνουν τις ζωές μας με πολλούς τρόπους αλλά με την πείρα της δικής μου ε, υπηρεσίας και ένωσης τα τελευταία 20 χρόνια και κυρίως 10 και αφού βοηθήσαμε ε, αρχές υπεύθυνες για την εξαγωγή των εκλογών και άλλους ενδιαφερομένους Είδαμε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να ενταχθεί η τεχνολογία στην εκλογική διαδικασία. Οι περισσότερε καλέ πρακτικέ, τι πρακτικέ, αναφέρθηκαν ήδη. Υπάρχουν και σχετικέ μελέτε, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα προβλήματα λύνονται και ότι η λύση ταιριάζει στι ανάγκε ε, αυτού που την αναζητά. Πρέπει να υπάρχει διαδικασία χάραξης της πολιτικής που να βασίζεται σε διάλογο, να συμμετέχουν όλοι, οι δικοί του χώρου, οι πολιτικοί δίνοντες, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, οι πολιτικοί. Θα πρέπει επίσης να είναι διαφανής και ανοιχτή η διαδικασία των προμηθεών το είπαν και ένα-δυο μιλητέ. Και τέλο, η σταδιακή υιοθέτηση με τις δοκιμές, την ε, εκπαίδευση σε αυτή τη διαδικασία και την σταδιακή εφαρμογή. Είναι λίγα τα μέρη όπου όλες αυτές οι φάσεις της διαδικασίας έχουν ακολουθηθεί σωστά, όμως ε, το λέμε ξεκάθαρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις όλα αυτά συμβαίνουν έστω και εκτός των εκλογών. Νομίζω λοιπόν η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι πώς η παρατήρηση των εκλογών διεθνώς μπορεί να προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει τι εκλογές αυτές. Δεν είναι κάτι που αφορά μία μόνο διαδικασία εκλογών, αλλά αφορά μία στις δύο περιπτώσεις και εκεί σίγουρα θα υπάρχει και χρήση και συζήτηση για τα τεχνολογικά μέσα. Ευχαριστούμε. Ξαβιέ Μελόν, ε, ανεξάρτητος ειδικό για θέματα εκλογών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφέρατε κυρίως τις απειλές και τους κινδύνους από τις τεχνολογίες κατά των διαδικασιών των εκλογών. Εάν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να αναπτύξετε λίγο το τι θετικά στοιχεία και φιλοδοξίες μπορούν να μας επιτρέψουν να επιδιώξουμε τα νέα τεχνολογικά μέσα στη διαδικασία των εκλογών. Δηλαδή, η, τα τεχνολογικά μέσα, ιδίως τα κοινωνικά δίκτυα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διεθνείς παρατηρητές εκλογών ως ε, εργαλείο για να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κ. Μικαλ Ευχαριστώ. Πρέπει να είμαι το 199, έτσι. Ναι. Ε, μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα υπόθηκαν αλλά νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των εκλογών, των αρχών που είναι υπεύθυνε για τι εκλογέ, ακούω τον εαυτό μου, πω, πω, ε, και τη πληροφορική. Πολύ ενοχλητικό. Και η άλλη ερώτηση είναι για τα κοινωνικά δίκτυα ε, και αυτό συζητιέται πολύ δημοσίω. Υπάρχουν διαφορετικά ζητήματα πληροφορική εκεί. Πρώτα απ' όλα οι αρχέ και πώ χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Ξέρουμε τι δυσκολίε τη ηλεκτρονική ψήφου κτλ. Αλλά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν περισσότερο να κάνουν με τον διάλογο των δημόσιο. Αυτό που εντάσσεται στην παραδοσιακή ίσω παρατήρηση μέσων μαζική ενημέρωση. Είναι δύο διαφορετικέ κατευθύνσει, δύο διαφορετικέ οδοί. Εκεί που έχουν κάτι κοινό βέβαια ότι οι παρατηρητές των εκλογών θα πρέπει να έχουν περισσότερες γνώσεις, ειδικέ γνώσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι εμπειρογνώμονες στις ε, αποστολές για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Εάν μιλάμε για μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα, είναι σαφώς ένας νέος ισχυρός παράγοντας στις εκλογικές διαδικασίες. Υπάρχουν πλατφόρμες και εταιρείε που παρέχουν κοινωνικά δίκτυα ως πολλές φορές δέχονται επικρίσεις ότι δεν, ε, και έχουν δεσμευτεί ότι θα βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους, αλλά δεν έχουν ακριβώς λογοδοτήσει. Αν το Facebook μας λέει ότι από εδώ και μπρο θα ε, έχω μόνο ε, δημόσια ανταλλαγή δεδομένων και κάτι τίποτα το κρυφό, αυτό πώς μπορεί κανείς να ξέρει αν θα υλοποιηθεί πλήρως βάσει των συστάσεων που έγιναν. Όλες αυτές λοιπόν οι ιστορίες θα πρέπει να μπορούν να λογοδοτούν ε, εφόσον μπορούν να βελτιώσουν το πλαίσιο της παρατήρησης. Και μετά για την πραγματικότητα του πράγματος μπορεί κανείς να παρατηρεί το χώρο των κοινωνικών δικτύων. Όπως είπε ο κ. Μελό, δεν μπορούμε τώρα να εφεύρουμε κάτι. Μπορούμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι παρατηρητέ, οι διεθνεί παρατηρητέ που έχουν ε, στραφεί σε διαφορετικέ πτυχέ του θέματο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει εδώ ένα σημαντικό ρόλο, διότι δεν έχουμε μόνο την παρατήρηση των εκλογών, αλλά και άλλα στοιχεία, όπω ε, το civic tech, την, στήριξη στην κοινωνία των πολιτών. Εδώ πρέπει να υπάρχουν τέτοια συστήματα που οι κοινωνίε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τι σχετικέ απειλέ. Όμω, για το δικό μας το θέμα, την παρατήρηση των ε, εκλογών, θα πρέπει να αποκτήσουμε τι ειδικέ γνώσει, να καταλάβουμε τι ακριβώ γίνεται. Γιατί σε μερικά χρόνια ο κόσμο θα έρχεται και θα μα λέει: Άκουσα ότι υπήρχε παρεμβολή της Ρωσίας στις εκλογές. Ε, έτσι είναι. Θα χάσουμε ένα μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας μας, εάν δεν έχουμε την απαραίτητη γνωμοσύνη για να μπορούμε Τουλάχιστον να ξέρουμε πώ συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίε. Είναι σημαντικό αυτό για τι διεθνεί παρατηρήσει εκλογών. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Και τώρα η Μάρκαρτ Καμά στο 106, βουλευτής από την Κένια. Άλλη μια βουλευτής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ομιλητές πολύ καλή πληροφόρηση. Επειδή είμαι από την Κένια, είχα πολλά ερωτηματικά και εγώ και βρήκα μερικές απαντήσεις. Ο ΠΑΤ έθεσε πολλά ζητήματα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι κατέρευσε η τεχνολογία. Η πολιτική κατέρευσε και απέτυχε. Ή κάποιοι από εμά σε κάποιο βαθμό. Τι θα γίνει όμως στις μελλοντικέ εκλογές. Τι θα πρέπει να κάνει. Τα δύο πρώτα που πρέπει να κάνει αμέσως η Κένια ποια είναι στη χρήση της πληροφορικής. Είπε ο συνάδελφος, ορισμένοι από εμά θεωρούσαμε ότι θα βοηθούσε το ηλεκτρονικό σύστημα. Στη συνέχεια, Σημείωσα ότι οι πολίτες πρέπει να κάνουν περισσότερα από ό,τι αυτή τη στιγμή. Να έχουν την ευκαιρία δηλαδή από τώρα, από την αρχή, να συμμετέχουν στην διαδικασία. Μήπως πρέπει να περιμένουμε λίγο. Γιατί εγώ, εγώ είμαι γερουσιαστής στην Κένια. Και περιμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να ε, επαληθεύσουμε τους εκλογικούς καταλόγους. Ήταν η μόνη δυνατότητα που είχαμε. Αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν ε, σε πολλά εκλογικά τμήματα. Και στη δική μου εκλογική περιφέρεια, σε κάποια εκλογικά τμήματα δεν λειτουργούσαν καν τα μηχανήματα. Ποιος στέει τώρα, η γαλλική εταιρεία που έκανε ηλεκτρονικά τις εκλογές, σε ποιον διαμαρτυρηθούμε. Συνεχίζω για το μέλλον των Διεθνών Αποστολών παρατήρηση Εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου πήραν οι παρατηρητές συνέντευξη το 2013 και την περασμένη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μόνη της ε, στην πάρτι εκλογών. Έχουμε αυτή τη συνεργασία που λέγεται ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργάζεται με τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού. Γιατί το λέω. Γιατί σε κάποιες αποστολές ευαίσθητες θα ήταν ίσως καλύτερο για μας αν συμμετείχαμε κι εμείς όχι εγώ στην Κένια, αλλά ίσω στην Ουγγάντα ή στην Τανζανία ή κάποιοι από την Ουγγάντα και την Τανζανία να παρατηρούν τις εκλογές. Γιατί μιλήσατε για δημιουργία ικανοτήτων και προβλήματα διαφάνειας. Ε, διαφάνεια ω προς τι και απέναντι σε ποιον. Είμαστε εκτεθειμένοι και σε ποιον. Και τελευταία ερώτηση. μετά ε, την ολοκλήρωση της αποστολής παρατήρησης των εκλογών. Σας ερωτώ, ως γερουσιαστής από την Κένια, σε ποιον παραδίδετε τα πορίσματά σας και τα αποτελέσματα. Τα λέτε στους Κενιάτες αυτά που παρατηρήσατε. Κάποια στιγμή είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ήταν εντάξει. Μετά ήρθε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και μπερδευτήκαμε. Πού την υποβάλλεται αυτή την έκθεση και εμείς πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση για να βελτιωθούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Έχω άλλες τρεις ερωτήσεις και μετά θα ζητήσω από τους ομιλητές να... Ε, εξαρτούντες να είναι σύντομοι για να μπορέσουν να απαντήσουν και τα μέλη του πάνελ, γιατί έγιναν πολλές ερωτήσεις. 188 θέση. Μένσον Ολουμπού από το Ίδρυμα Κλίντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τα μέλη του πάνελ για τη συνεισφορά τους. Εγώ είμαι από την Ιγυρία, όπου είχαμε εκλογές το Φεβρουάριο μάλλον θα έχουμε το Φεβρουάριο του 2019. Έχουμε 80 εκατομμύρια κατοίκους. 84 ε, εκατομμύρια και στην Αμπούτζα ε, είναι η Κεντρική Φορευτική Επιτροπή και 91 πολιτικά κόμματα. Καλά τα δύο είναι τα βασικά. Πρόσφατα σε μια εκτίμηση που έγινε από τα δικαστήρια είδαμε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα κηρύγματα μίσους μπορεί να πυροδοτήσουν τη βία. Συνεργαζόμαστε με διάφορους ε, εταίρους για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κηρύγματα μίσους και τα fake news, τις ψευδείς ειδήσεις. Και τα social media λοιπόν είναι στοιχείο της εκλογικής παρατήρησης. Πρόσφατα εγκρίθηκε ένας νόμος για να προστατεύει την νεολαία υπάρχουν κάποια πολύ υψηλά τέλη για να καταθέσει κανείς την υποψηφιότητά του και πολλοί νέοι που ενδιαφέρονται και για τα δύο ισχυρότερα κόμματα δεν μπορούν να το κάνουν λόγω κόστους. Ως ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, εμείς πώς θα εξασφαλίσουμε να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί τους τα όσα λέμε. Γιατί όταν μιλάνε οι διεθνείς παρατηρητές αγωνιούν να ακούσουν τι θα πούν οι εκάστοτε κυβερνήσει και τους παρακολουθούν. Αλλά όταν εμείς που είμαστε από την ίδια χώρα εκφράζουμε κάποιες απόψεις, δεν μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Είναι σημαντικό να το θέσουμε και εδώ γι' αυτό. Και το 2019 είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία για την Νιγηρία και είναι πρώτη φορά που η τρέχουσα κυβέρνηση διοργανώνει γενικές εκλογές. Στο παρελθόν είχαν ε, διοργανώσει περιφερειακές εκλογές με επιτυχίες και αποτυχίες. Το σημαντικό είναι οι γενικές εκλογές το Φεβρουάριο να είναι ελεύθερες, αξιόπιστες και να εκφραστεί η λαϊκή βούληση και η λαϊκή ετοιμιγορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος και τελευταίος. Ελπίζω να το πω σωστά, διότι δεν διαβάζω πολύ καλά το γραφικό χαρακτήρα. Μοχάμετ Φάκη Βίνι Φάτζι. από το Κοινοβούλιο της Κένιας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όσους μίλησαν από το πάνελ, κυρίως για το θέμα της Κένιας. Ήθελα πολλά να, να πω, αλλά έχω ήδη καλυφθεί. Ένα είναι το βασικό. Όταν μιλάμε για έναν κρατικό φορέα, όπως την ABC στην ε, Κένια, την Ανεξάρτητη Φορευτική Κεντρική Επιτροπή, πώς μπορεί κανείς να εξορροπήσει το κρατικό συμφέρον και το ιδιωτικό συμφέρον μιας εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει να συγκεντρώσει πληροφορίες για μια εκλογική διαδικασία η οποία γίνεται για το δημόσιο συμφέρον. Επίσης στην Κένια ε, υπήρξε μια επιτυχής προσπάθεια των ε, υπευθύνων των παρατηρητών να δουν τι πρόβλημα υπήρξε με τα ψηφιακά και την ατυφή την εταιρεία που είχε αναλάβει το σύστημα και παρόλο που υπήρξε ένταλμα από τα ανώτατα δικαστήριο να δώσουν τις απαντομένε πληροφορίε, η εταιρεία αυτή η ιδιωτική, δεν ε, μπόρεσε να γίνει κατά τέτοιο λόγω αντίστασή τους. Τελευταίος ομιλητή ο Έστεν Ταουία, από το Κέντρο για την Ισότητα των φιλων Στη θέση 81, συγγνώμη. Ευχαριστώ, είμαι από την Γκάνα. Λοιπόν. Από το 2000 η συμμετοχή της προφορικής της εκλογές αυξάνεται. Αλλά... Αλλά δεν ξέρω τώρα αν είναι τα συμβόλαια που υπογράφουμε ή τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Αλλά τις περισσότερες φορές αυτό αποκλείει πολλούς πολίτες. Διότι πας στο εκλογικό τμήμα και δεν δουλεύουν τα μηχανήματα σου λένε πήγαινε πριν τα χέρια σου ξανά έλα, έλα αργότερα. Χρειαζόμαστε κάποια μηχανήματα, κάποια πληροφορική που να δουλεύει. Τι μας συστήνεται. Κοιτάξτε, πολλές, την περισσότερες φορές ε, τα εκλογικά τμήματα είναι ανοιχτοί χώροι, όπως είναι εδώ στην Ευρώπη. Που δεν είναι όπως είναι εδώ στην Ευρώπη που είναι κλειστή. και για τα κοινωνικά μέσα. Οι οργανισμοί διαχείρισης των εκλογών δεν ξέρουν τι γίνεται με τα κοινωνικά μέσα. Δεν μπορούν να εντοπίσουν τις ψεύτικες ειδήσει για τα αποτελέσματα, για παράδειγμα. Υπάρχει τρόπος που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να τους βοηθήσει με κάποια μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Γιατί είναι πολύ σοβαρά. Κάτι άλλο επίσης για την Κένια. Γίνεται hacking πολλές φορές. Ποιος παρακολουθεί ποιον, αυτό είναι το θέμα. Και πώς καταλαβαίνεις ε, αν έχουν μπει στα συστήματά σου. Δεν ξέρω τώρα τι λύση μπορούμε να βρούμε, γιατί στην Κένια ήταν μεγάλο θέμα. Και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης είναι ότι κάποιοι μπήκαν μέσα και άλλαξαν τα αποτελέσματα. Και είπαν ότι γι' αυτό το λόγο υπήρξε νοθεία. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Συγγνώμη. Δεν έλαβα το χαρτί σας ότι θέλατε το λόγο. Αλλά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Φάτμα Τζαντζάρα Ντεμπελέ από το Μαλί, από τον Πόλο Παρατήρησης των Πολιτών. Θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, ασφάλεια και, τις ε, και την ειρήνη. Μήπως αυτό σημαίνει ότι πάντα οι παρατηρητές ενώ δεν ε, βλέπουν τι έγινε, επειδή δεν μπορούν ε, να μπουν στα στοιχεία προφορικής, είναι υποχρεωμένοι παρόλα αυτά να δώσουν μια γνώμη. Ακόμη και αν δεν έχουν δεδομένα που να τους επιτρέπουν να πιστοποιήσουν τι έχει γίνει για τις εκλογές. Επειδή πάνε σε πολύ λίγα εκλογικά τμήματα και είναι δύσκολο να πάνε. Διότι έχουν μεγάλη αξιοπιστία οι διεθνείς παρατηρητές έναντι των κομμάτων και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και στην κοινή γνώμη. Άρα έχει στρατηγική σημασία η γνώμη που θα δώσετε για το αν θα γίνουν αποδεκτά τα αποτελέσματα και για το εάν θα προκύψουν κατόπιν συγκρούσεις. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Εάν ακυρώσει η δικαστική εξουσία κάποιε εκλογές μετά την ε, θετική σα Τι στάση έχετε. Και τρίτον, ο τελευταίο ομιλητή είπε ότι πρέπει να ενημερώνεται το εκλογικό σώμα. Είπε ότι οι εκλογικέ δεν μπορεί να είναι αποκομμένες από την καθημερινή πολιτική και κοινωνική ζωή. Πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση. Αλλά στις χώρες μας μόνο 20% του πληθυσμού έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση. Τι συστήνεται. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που δώσατε το λόγο και την κατανοήσή σας. Ευχαριστώ κυρία μου. Λοιπόν, στρέφομαι προς τους ε, ομιλητές μας. Ποιος θέλει το λόγο να ξεκινήσει πρώτος. Έχουμε πολλέ ερωτήσεις. Τάνια, ξεκινήσει εσύ. Θα προσπαθήσω. Δεν θα απαντήσω στις ερωτήσεις που είχαν άμεση σχέση με τις παρατηρήσεις εκλογών ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ξέρεις μία που τη βρήκα ενδιαφέρουσα. Όταν ρωτήσατε εάν η παρατήρηση των εκλογών πρέπει να είναι πάντα μόνο σήμαντη προς μία κατεύθυνση. Εγώ έχω ε, βρεθεί στην Αφρική πολλές φορές ε, ως ε, παρατηρητής εκλογών και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τελευταία χρόνια για τον ΟΝΤΙΡ του ΟΑΣΕ και για μένα ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι το εξή. Η παρατήρηση των εκλογών στον ΟΑΣΕ είναι κάτι που βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Είναι μια συμφωνία όπου συμμετέχουν όλα τα συμβαλόμενα μέρη, ότι θα ανοίξουν τις χώρες τους για να γίνει η παρατήρηση εκλογών. Και ανέφερα δύο χώρες, την Εσθονία και τις Ηνωμένε Πολιτείες, όπου έχω συμμετάσχει σε παρατήρηση εκλογών. Και αυτό είναι μία από τις μεγάλες ε, έτσι, ε, τα μεγάλα του μάλλον ε, αυτή η αμοιβαιότητα. Οπότε Ε, ήταν πολύ καλό αυτό που προτείνατε, νομίζω κάποιος από την Κένια, ότι θα είναι πολύ εμπλωτιστικό αυτό και για την εμπειρία των παρατηρητών από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε μια αναφορά στην προσαρμογή ε, του τρόπου με τον οποίο γίνεται η παρατήρηση των εκλογών, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ε, της υλοποίησης των νέων τεχνολογιών. επειδή υπάρχουν στοιχεία μακροπρόθεσμα ε, γιατί αυτά είναι κάτι που χρειάζονται σχεδιασμό εκ των προτέρων, ιδιαίτερα υπογραφές των συμβολέων και, των, και προκήρυξη των διαγωνισμών. Ε, είναι κάποια στοιχεία που θα πρέπει να υλοποιούνται ε, νωρίτερα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, πολλοί. Θα ήθελα να πω κάτι για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αναφέρθηκα σε αυτό προηγουμένως. Δεν έχουμε μεθοδολογία εδώ. Ε, βέβαια, είναι ένα τμήμα των αποστολών παρατήρησης και είμαστε στο, στο στάδιο τώρα του πειραματισμού. Θα πρέπει να μπούμε όμως προς τον ορισμό για το πώς ορίζονται τα social media, η κοινωνική δικτύωση και σωσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Οι τεχνολογικές εταιρείες οι ίδιες δεν θέλουν τον εαυτό τους μέσα ενημέρωσης, media. Λέει ανταλλάσσουμε πληροφορίες και μεταξύ αυτών είναι και ε, ε, τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό ισχύει ε, μέρη μόνο διότι έχουν ε, δημιουργήσει και εφαρμογές για δημοσιεύσει, αλλά επιλέγουν και όλα τα μέσα ενημέρωσης τα οποία θα απευθύνονται στου χρήστες τους. Δηλαδή είναι και εκδότε οι ίδιοι. Ε, δεν τους θεωρούμε αποκλειστικά όμως μέσα, αλλά τους θεωρούμε ε, εργαλεία προεκλογικής εκστρατείας. Και είναι πολύ σημαντικό εδώ να το λαμβάνει υπόψη της αποστολή παρατήρησης. Αυτό το κάνουν και αναλυτές του τύπου, αλλά και πολιτικοί αναλυτές. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε και γνώση των τοπικών μέσων ενημέρωσης και παρατηρητές να το κάνουν αυτό. Ε, ε όχι μόνο τα μέσα ενημέρωση, αλλά και την εκτίμηση κάποιων πανεπιστημιακών από τη χώρα στην οποία γίνεται η παρατηρήση εκλογών. Εγώ είμαι από την Ιταλία και ε, επικράτησε η άποψη ότι στις τελευταίες εκλογές έπαιξαν τεράστιο ρόλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εμπειρικές μεθόδους όπου μετρούσαν την θεαματικότητα και ε, ε, κατέληξαν ε, στο συμπέρασμα ότι δεν ίσχυε αυτό, ότι το, τα, τα, όσα έλεγαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσαν και στα βασικά μέσα ενημέρωσης και ο κόσμος ενημερωνόταν κυρίως από τη τηλεόραση. Και ένα τελευταίο. Όταν με προσκάλεσαν να έρθω στο πάνελ εδώ, η Επίτροπος Γκάμπριελ ήταν μία από τις συμμετέχουσες. Και μάλιστα με ενδιαφέρε πάρα πολύ γιατί και άκουσα και την ε, σημερινή της ομιλία. Και ένα από τα ενδιαφέροντα είναι ότι τώρα παρατηρώ μια χώρα που βάζει πολύ ψηλά στο σύνταγμά της την ελευθερία της έκφρασης. Δηλαδή ακόμα και η χρηματοδότηση των ε, προεκλογικών ε, εκστρατιών είναι τελείως αρρύθμιστη γιατί θεωρείται ελευθερία της έκφρασης ιερή. Στην Ευρώπη το κοινοβούλιο σας έχει προχωρήσει με διαφορετικό τρόπο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και όπως είπα και προηγουμένως, το ανέφερε και η Επίτροπος Γκάμπριελ στην ομιλία της, ε, υπάρχει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό και αυτό είχε αντικτυπώ πολύ πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων και έχει γίνει και ορόσημο και πολύ υψηλά πρότυπα και επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές εταιρείες ε, λειτουργούν και δραστηριοποιούνται πολύ πιο πέρα από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κινηθεί προς νέα κατεύθυνση, το είπε και η προς τη διαφάνεια, στους αλγορίθμους, διαφάνεια στη ροή των διαφημίσεων στο διαδίκτυο και περιμένουμε ενδιαφέρον ε, όλα αυτά. Και ήδη επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εταιριών τεχνολογίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλες εταιρείες ήδη Ε, βάζουν σε βάσεις δεδομένων όπου υπάρχει δημόσια πρόσβαση ε, τις δαπάνες τους για διαφήμιση και άλλα τέτοια στοιχεία. Αυτά είναι πρωτοφανή. Και αυτό μάλλον επηρεάζεται από τις νομοθετικές προσπάθειες που συνεχίζονται στην Ευρώπη. για μένα η συνεδρίαση η σημερινή είναι πάρα πολύ σημαντική και από αυτή την έννοια. Ιδιαίτερα ακριβώς αυτή τη στιγμή που έχω ε, ένα πόδι στην Ευρώπη και ένα στην Αμερική. Για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τρόπο επικοδομητικό. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρίτια. Πρέπει να φύγω ε, μόλις τελειώσω γιατί έχω κάποιες υποχρεώσεις. Αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο περισσότερες ερωτήσεις γίνεται. Αλλά είναι πάρα πολλές. Πολλές έχουν να κάνουν με το τι μπορεί να κάνουν οι αποστολές. Είναι σημαντικό λοιπόν. Και για να είμαι σύντομη, ενθαρρύνω όσους ε, ενδιαφέρονται να ε, δουν τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει η Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι η αποστολή μας είναι να δούμε σε τι βαθμό οι εκλογές στην πράξη ανταποκρίνονται στην εκλογική νομοθεσία. Ε, αν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ε, εκλογέων, με βάση ακριβώς την νομοθεσία. Με βάση τους νόμους και τις παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε συστάσεις και αυτό κάνουμε. Όσοι ενδιαφέρονται για τα διδάγματα από την Κένια, δείτε τι ακριβώς είπαμε, γιατί υπήρξε πολλή επίκριση σε μια αρχική έκθεση που δεν αναφέρθηκε στον τύπο, αλλά όπου βλέπετε τις λεπτομέρειες της δουλειάς μας και για συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, αυτή η ισχυρισμοί ότι υπήρξε hacking που μας είπε η αντιπολίτευση μας έδωσαν και στοιχεία που μας έλεγαν πως ήταν ενδείξεις και τις εξέτασαν διάφοροι εμπειρογνώμονες ε, πολύ γνωστοί κυβερνοασφάλειας και δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ήταν hacking. Αυτό δεν αποδεικνύει πως δεν υπήρξε hacking, αλλά δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Και διάφοροι εμπειρογνώμονες για τέτοια θέματα συμφώνησαν πως δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Αυτό ίσως οδήγησε σε περισσότερη πόλωση, αλλά το εξετάσαμε όσο μπορούσαμε, όπως και άλλοι, και δεν βρήκαμε να υπάρχουν στοιχεία σε αυτά τα log του ίντερνετ. Μετά... Δαρία. Ε, ρώτησε κάποιος για την Κεντρική Φορευτική Επιτροπή στην Γένεια και στις 16 Αυγούστου ε, πιέσαμε να υπάρχει διαφάνεια στα ε, έντυπα. Και θεωρώ πολύ σημαντικό ότι οι δημόσιοι θεσμοί όπως κεντρικές εφορευτικές επιτροπές αλλά και κυβερνητικά ε, όργανα είναι αυτοί που λογοδοτούν. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη δημόσια λογοδοσία, ακόμα και όταν είναι ιδιωτικές οι εταιρείε που ενέχονται. Και τι σημαίνει αυτό, αποφυγή της διαφθοράς, ε, βελτιστοποίηση των μηχανισμών ε, λογοδοσίας και στην ανάθεση των έργων και στην υπογραφή των συμβάσεων. Και ιδιαίτερα ε, με την πληροφορική ε, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν οι εταιρείε. Πού καταλήξαμε στην Κένια λοιπόν, ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την εμπιστοσύνη και όλοι ρωτήσαμε τι να κάνω, ρωτήσατε εσείς, να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε τη τεχνολογία ή να ψηφίζουμε με χαρτί. Εγώ δεν έχω πρόβλημα ε, με το μέσο που ή το υπόστρωμα που χρησιμοποιείτε αν είναι χαρτί, αν είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητες επαληθεύσεις, να ελέγχεται ο ελεγκτής. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι χαρτί ή ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το θέμα είναι να γίνονται πολλές επαληθεύσεις και να υπάρχουν πολλές μέθοδοι έτσι ώστε αν ε, καταρρεύσει μία αποτύχη να περάσουμε στην επόμενη να υπάρχουν έλεγχοι και αντίβαρα ε, σε αυτά τα συστήματα. Και πάρα πολύ γρήγορα για την ελευθερία της έκφρασης και το ε, πλήθοπορισμό και την παρατήρηση από πολίτες που συλλέγουν ε, χρήματα. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει η ελευθερία της έκφρασης για τα bot, δηλαδή ένα άτομο θα πρέπει πάντα να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Αυτό είναι πολύ σημαντική αρχή. Αλλά ένα bot, ένα αυτόματος, ένας αυτόματος λογαριασμός σε υπολογιστή έχει ελευθερία έκφρασης. Οι τεχνολογίες ε, προχωράνε συνέχεια. Τώρα είναι δυνατές και βαθιές ψευδείς ειδήσει. Είναι δυνατόν να φτιάξει ένα βίντεο που να λέει κάποιος, να εμφανίζεται κάποιος να λέει κάτι που δεν το έχει πει ποτέ και ένας απλός άνθρωπος ε, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Εγώ έχω δει φωτογραφίες παραποιημένες, έγραφα παραποιημένα. Κάθε είδος ε, παραποιημένες, ε, παραποιημένους ισχυρισμούς που μας τους φέρνουν και μας λένε βεβαίως να εδώ υπήρξε βία, υπήρξε κακή συμπεριφορά και εμείς καταλήξαμε ότι αυτές οι εικόνες ή αυτά τα αποσταρίσματα στη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν παραποιημένα τι είναι όταν λέμε ότι το πλήθος μπορεί να βοηθήσει, ποιο είναι το πλήθος, μήπως είναι bot, μήπως το πλήθος μπορεί και αυτό να, ε, να, να προωθήσει ψευδείς ειδήσει και να παρεποιήσει ειδήσει. Έχουμε πολλές αποστολές και η Αφρικανική Ένωση είναι σημαντική και άλλοι στέλνουν παρατηρητές και είναι πολύ σημαντικό υπάρχουν και επιτόπου παρατηρητές. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Είναι διαφόρων ειδών αυτοί οι παρατηρητές. Αλλά αν υπάρξει διαφάνεια θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την αλήθεια. Και καταλήγω όπως ξεκίνησα, καμία αποστολή μπορεί να δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Μπορούμε να αξιολογήσουμε το πώς γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα, αλλά δεν υπάρχει πραγματικά εμπιστοσύνη, καμία τεχνόλογη, κανένα ιδιαίτερα περίπλοκο και προηγμένο σύστημα δεν θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε τη βέλτιστη διαφάνεια, τι βέλτιστε δυνατότητε επαλήθευση και ελέγχου. Μόνο έτσι θα επανέλθει αν έχει καταργηθεί η διαφάνεια. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Μαρίτια. Έχουμε ξεπεράσει αρκετά το χρόνο μας. Σε 4 λεπτά, 18 και 40, θα χάσουμε τη διερμηνία. το συγγνώμη γι' αυτό. Παρακαλώ να δείξετε κατανόηση. Θα ολοκληρώσουμε το πάνελ όπως μπορούμε μετά τις 18 και 40. Ήδη έχεις το λόγο. Ευχαριστώ για αυτή την πρόκληση, όχι μόνο χρονική πίεση, αλλά είμαστε τα τελευταία εμπόδια πριν το κοκτέιλ εμείς. Θα προσπαθήσω λοιπόν γι' αυτό να είμαι σύντομος. Και να μην επαναλάβω πράγματα που ήδη πώς θα δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα ε, εκλογικών διαδικασιών που να βασίζονται στο, στο ψηφιακά μέσα. Θα δείτε στις μελέτες 5-6 μελ... συστάσεις που είναι σημαντικές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι μέρος της συνολικής αναθεώρησης της κατάστασης των ε, ψηφιακών συστημάτων και να μην το δούμε ως κάτι το μονομένο. Δύο, να είναι το δυνατόν ευρύτερος ο δημόσιος διάλογος για να ε, αναλάβει την ευθύνη των ελέγχων που θα γίνουν η ίδια κοινή γνώμη. Τρία, άμεση πόρια του δύο, ε, μέγιστη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, των προμηθειών και το καθεξής, της ανάθεσης. Τέσσερα, ένα χρονικό πλαίσιο, χρονοδιάγραμμα, το οποίο να μπορεί κανείς να το διαχειριστεί. Μην περιμένει να γίνει σε χώρες που δεν έχουν εισάγει ακόμα τα μηχανήματα και δεν είναι αξιόπιστες εκλογέ. ή να έχουν αγοραστεί εγκαίρω και να μην είναι πολύ κοντά σε εκλογέ ή αγορέ, α πούμε, γιατί δεν εμπιστεύονται τα νέα μηχανήματα οι άνθρωποι. Και πέντε, ε, νομοθεσία που από την αρχή να προβλέπει τακτική ε, αναθεώρηση, αξιολόγηση που να έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Δεύτερη παρατήρηση. Και... Και το λέω ευλογώντας τα γένια μου λίγο αυτό. Εδώ θέλουμε ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ε, για την εκπαίδευση, για τους ανθρώπους που εργάζονται στην ε, Επιτροπή της Βενετίας, που παρακολουθούν εκλογικές διαδικασίες. θα πρέπει να μην χρηματοδοτούνται από εταιρείε που έχουν άλλε προτεραιότητε από το δημόσιο συμφέρον αυτέ οι οδέσει, οι καταρτήσει. Είναι σημαντικό η εκπαίδευση ε, στο σχεδιασμό τη ε, να γίνεται με έναν τρόπο επιτυχή. Ξέρετε το λεγόμενο bridge training όπως είχε ονομαστεί. Ε, ήταν πολύ επιτυχημένο, το ίδιο και για τις πλατφόρμες. Μπορεί κανείς λοιπόν να σχεδιάσει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και πολλές σωστέ επενδύσεις να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τρίτη παρατήρηση για το τι μας λένε οι ακαδημαϊκές μελέτες και τα στοιχεία. Ε, για όσο περισσότερο εξοπλισμένη είναι η Εφορευτική Επιτροπή, τόσο καλύτερα και τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή, η σωστή δίκτυα συγκριτικής αξιολόγησης και ε, σωστή μέτρηση των στοιχείων και σωστές παρατηρήσεις και οι χώρες ε, μπορούν να κάνουν πολλά για την παρατήρηση των εκλογών. Θα ήθελα κάτι να πω και για τις ψευδές ειδήσει και τα μπότα, αλλά δεν ε, θέλω να φάω χρόνο από το συνάδελφο. Ευχαριστώ. Uh, Τελευταίος, ο Πατ Ζητώ συγγνώμη που δεν σιωπώ με κίνδυνο να εκτεθώ ε, από κάποια πράγματα που λέω. Όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος, με βάση την συμφωνία με την γραμματεία, η διερμηνία θα διακοπεί τώρα. If there is an election in which the people do not trust, it will not be accepted. If there is an election in which the competitors do not trust, they won't take the outcome. The consequences of these